Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω στην κοινή συνεδρίαση Envy Affet. Ε, χαιρετίζω λοιπόν ιδιαίτερα όλους τους συναδέλφους από την Envy. Περνάμε στο σημείο 1 της ημέρησιας διάταξης. Παρακαλώ. Έγκριση της ημέρησιας διάταξης. Κύριε Πρέντα, έχετε αντιρρήσει ω προς την ημερήσια διάταξη. Όχι. Ωραία. Εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Ωραία. Οπότε, έγκριση πρακτικών. Εντάξει. Ωραία. Οπότε, περνάμε στο σημείο 3. Κλιματική διπλωματία. Έχουμε μια έκθεση. Αν Λίτς και Λάιν ήταν οι συγητές μας.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 Πώς είμαστε? Λοιπόν, 98% ψήφισαν, πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται.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 Δεκτή. 106 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχέ Δεκτή. 109 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά αποχέ Απορρίπτεται.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 Θέλετε να ελέγξουμε το 131. Να ελέγξουμε το 131. The vote is... Πέρας. So, Απορρίπτεται. Καλώς. «132 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 134 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε 134. Πέρας.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 Πέρας. Δεκτή, αλλά με πολλές αποχές. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας.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 Αποχές. Να την ελέγξουμε. Την 200. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 201 και 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές.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 Πέρας. Εγκρίνεται. 2.28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ελέγχονται 2.25. Μα την ψηφίσαμε. Καλά. 2.25 έκανα λάθο. Λοιπόν, 2.25 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. 2.26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 Πέρα τη φοφορία και απορρίφθηκε. 4 και 5 τη ψηφίσμου μαζί υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτονται. 6 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 9 υπέρ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 αποχές. Θα ελέγξουμε για τις 42 και 43. Ψηφίσατε όλοι, πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές,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 Δύο ακόμα πρέπει να ψηφίσουν. Δεν θέλετε να συμμετάσχετε. Άλλος ένας. Ακόμα. Ωραία. Πέρα της ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκε 90 ψήφοι υπέρ, 19 κατά και δύο αποχές. Συγχαρητήρια στους συζητητέ. Οπότε ολοκληρώθηκε εδώ η κοινή μας συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ στους συναδέρφους της Επιτροπής Περιβάλλοντος που ήρθαν για την ψηφοφορία εδώ.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 Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τώρα με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών. Νομίζω ότι επαναπρογραμματίστηκαν τα μηχανήματα, οπότε είμαστε στο σημείο 2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης πρώτα απ' όλα. Έχετε σχόλια μήπως? Ο κύριος Στροβίτσιος. Έχετε κάτι να πείτε κύριε Πρέντα. Ε, για τη Μολδαβία. Θέλετε να μας ενημερώσετε. Αν είναι αλήθεια αυτά που ακούσαμε, ε, ότι το δικαστήριο δεν συμφώνησε στο Κίσιους όσον αφορά την Αστάσια που εκλέχτηκε ως νέος δήμαρχος, ε, σίγουρα πρέπει να αντιδράσουμε και έγκαιρα. Ο Κρίστιαν Πρέντα, ήδη προηγουμένως στην κοινή συνεδρίαση που είχαμε με την ΕΝΒ, το ανέφερε και προσπαθούμε να πετύχουμε σήμερα να έρθει στην Επιτροπή μας κάποιος από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να μας ενημερώσει για το τι γίνεται ακριβώς στο Κίσινα. Και μόλις έχουμε νεότερα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα σας ενημερώσουμε. Ωραία. Κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί για λίγα λεπτά να αλλάξουμε την ε, ημερήσια διάταξη όπως καταλαβαίνετε για να μπορέσει να μπει το θέμα της Μολδαβίας αν έρθει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ωραία. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. αλλιώ σημείο 3, ανακοινώσεις της Προεδρίας. Δεν έχω τίποτα να πω. 4. Έγκριση των πρακτικών των ε, διάφορων συνεδριάσεων. 19 και 20 Μαρτίου, 12 Απριλίου, 17 Απριλίου και 26 Απριλίου. Σχόλια επί των πρακτικών. αν δεν υπάρχουν σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θεωρούνται εγκεκριμένα. Και ερχόμαστε τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σημείο 5. Συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ιράκ. Και σημείο 6. Συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ιράκ. Η συγγήτρια και για τα δύο αυτά θέματα είναι η κυρία Σαϊφή. Μήπως η κυρία Σαϊφή θέλει να πει κάτι, παρακαλώ. Α, όχι, δεν έχετε τίποτα να πείτε. Πολύ ωραία. Τότε περνάμε απευθείας στην ψηφοφορία. Και αρχίζουμε ψηφίζοντας το σχέδιο όσον αφορά την ε, σχέση και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και του Ιράκ από την άλλη. Είναι μια νέα ψηφοφορία, υπέρ παρακαλώ. Α, όχι, είναι ηλεκτρονικά ονομαστική ψηφοφορία, ναι. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 51 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Και τώρα Α, και η Νίνα Γκίλαρα, 52 υπέρ. Και τώρα ερχόμαστε στο κατάλογο ψηφοφορίας και αρχίζουμε με την τροπολογία 51. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 79 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Για τον αντιπρόεδρο το κάνουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 82 υπέρ. 83 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Να ελέγξουμε. Ωραία. 83, έτσι, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ.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 Συνολικά είμαστε 64 και ψηφίζουν 61. Άρα τρεις κοιμούνται. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 105 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, Την 105 θέλετε να ελέγξουμε. Ποια, την 105 θέλετε να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά. Ωραία. 105 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκε με σαφή πλειοψηφία. Ζητάτε να ελέγξουμε ενώ είναι τόσο σαφές το αποτέλεσμα. Εκτός μικροφώνου η παρέμβαση του βουλευτή δεν την ακούμε στην καμπίνα. Πρόεδρος, μα βλέπετε, το δείχνουν οι επικεφαλείς των ομάδων, οπότε ξέρουμε τελικά πώς θα ψηφίσουν τι. Συνεχίζεται η παρέμβαση εκτός μικροφώνου, δεν την ακούμε. Κύριε Φλέκενστάιν, παρακαλώ. Πρόεδρε, ο συνάδελφο σήμερα το πρωί είχε κάποιε δυσκολίε από ό,τι φαίνεται. να έρθει εδώ στην πρώτη σειρά. Θα βλέπετε καλύτερα, ξέρω εγώ. Πρόεδρο, συνεχίζουμε. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 113 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 121 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 122 κατά τμήματα, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Πρώτη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ένα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 5. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 20. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Και σαφώς απορρίφθηκε. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε για την 25 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε σαφώς. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33 σε δύο τμήματα ή όχι. Εγκρίναμε την 7, τη συμβαστική. Ναι, οπότε το πρώτο τμήμα καταπίπτει. Οπότε ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα μόνο, σωστά. Τρία, ε, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44 Θέλετε να ελέγξουμε. Καλώς. 42. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος της προφορίας. Απορρίφθηκε. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τη 46. Ψηφίστε. Πέρας της φοφορίας. Απορρίφθηκε. 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα ερχόμαστε στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, δεν θέλω να εντείνω τις γερμανοπολωνικές σχέσεις, λέει ο Πρόεδρο. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του τροποποιημένου σχεδίου έκθεσης. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Δύο ακόμα πρέπει να ψηφίσουν, παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 51 ψήφοι υπέρ, 3 κατά. Συγχαρητήρια κυρία Σαΐφη. We Να περάσουμε τώρα στο σημείο 7 σύσταση προ το Συμβούλιο σχετικά με την 73η Σύνοδο τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ε, Εισηγητή ο Όγκεν Φρόιντ. Θε να πει δύο λόγια, ε, Όγκεν, παρακαλώ. I was advised. Μου δόθηκε η συμβουλή να μην πω τίποτα. Παρ' όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητέ και συναδέλφου για την εκπόνηση αυτή τη έκθεση και ανυπομονώ για το τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ συνάδελφε. Η κυρία Λόχμπίλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια προφορική τροπολογία, διότι χθε το βράδυ η ΕΙΠΑ έφυγε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ε, προς υποστήριξη λοιπόν του συγκητή θα ήθελα να διαβάσω και το κείμενο της προφορικής τροπολογίας. Εκφράζει τη θλίψη για την απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν και να σταματήσουν να συμμετέχουν ε, στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΙΕ, γιατί είναι πολύ σημαντικό ο φορέα αυτό και καλούν τι ΗΠΑ να ανακαλέσουν την απόφαση αυτή. Στην έκθεσή μα επικρίνουμε ήδη τι διάφορε ελλείψει και παραλήψεις. Αυτό όμως, ε, επειδή είναι της τελευταίας στιγμής είδηση, ελπίζω να γίνει δεκτό τροπολογία. Πρόεδρος, δεν έχω εγώ κάποιο πρόβλημα. Σχόλια από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Μπορείτε να ανοίγετε και το μικροφωνό σας. Με συγχωρείτε, αλλά δεν κατάλαβα. Θέλετε το κείμενο να αντικαταστήσει κάτι κυρία Λόχπιλου. Είναι μια επικαιροποίηση του κειμένου, μια προσθήκη. Ήδη υπάρχουν επικριτικά σχόλια στο κείμενο, απλώς θέλουμε ε, ε, να αναφέρουμε και τις ε, παραλήψεις λόγω της δράσης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ναι, θα την ψηφίσουμε στο τέλος αυτήν την τροπολογία. Είναι μακροσκελής ο κατάλογος ψηφοφορίας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν Προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι για να κάνουμε και γρήγορα. Να ξεκινήσουμε με την τροπολογία 48 Τάνοκ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε την 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Μας λείπουν τρεις. Πέρας. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ελέγχουμε την 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 30 προς 27. Μικρή διαφορά. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 57. Πρέπει να ελέγξουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. 65 Κόβατσεφ. Ναι, μου ξέφυγε. Ε, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε για την 71 του κ. Λάιναν. Άρχεται η ψηφοφορία. Από ό,τι φαίνεται, οι τρει συνάδελφοι έχουν φύγει από την αίθουσα ή δεν του ενδιαφέρει να ψηφίσουν. Ενδιαφέρον αυτό. Πέρας. Απορρίφθηκε. 72 έως 75 ε, από κοινού ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 88 είναι τώρα. 88 υπέρ, κατά, αποχές, Έλεγχο. Ελέγχουμε για τον 88, άρχεται η ψηφοφορία. Οι τρει συνάδελφοι ακόμη είναι αποκοιμισμένοι. Πέρας, εγκρίθηκε. 89, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 90, υπέρ, κατά, αποχές, Έλεγχος. Ψηφίζουμε για την 90. Ε. Πέρας. Απορρίδεται. 91 έως 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 πίπτη. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 121. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 135 με προφορική τροπολογία. Συμβαστική 12 ζητάτε έλεγχο. Πολύ καλά. Μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε με μικρή διαφορά. 135 την προφορική τροπολογία 1, Κόφατσεφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 136. Θα είναι ακόμη μεγαλύτερη διαφορά πιστεύω. Μας λείπουν έξι συνάδελφοι. Ξυπνήστε παρακαλώ. Πέρας. 27 προς 30. Απορρίπτεται. 137. Κατά τμήματα. Σε δύο τμήματα. Πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 27 προς 25. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε για το δεύτερο τμήμα. Πέρας. Εγκρίθηκε. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά ελέγχουμε για την 140 Πέρος. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 145. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 146, κύριε Λάινεν του κυρίου Λάινεν. Πέρας. Απορρίφθηκε. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ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 Συμβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 179 Τάνοκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180-181. Από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 182. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 182. Τα κυρίας Μούντι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 183. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 184. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 185. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 186. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 187. Υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος για τον 187, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 193, Λοχμπίλερ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 193 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 194. Καταπίπτει. Ναι, εγκρίναμε την προηγούμενη. 196 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 198 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την 198. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίπτεται αλλά να ελέγξουμε 207 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. «24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται». «213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται». «214 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Θα βοηθούσε εάν σηκώνατε λίγο τα χέρια. Άρχεται η ψηφοφορία. Τρεις συνάδελφοι μας λείπουν ακόμα, αλλά η ψηφοφορία έληξε. 28 προς 24 εγκρίνεται. 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 218 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 219 υπέρ κατά αποχές 219 έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 222. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 223. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 225. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ή απορρίπτεται. 225 να ελέγξουμε του κυρίου Σόλτς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 234 σαϊφή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 236 διαγράφεται. 237 υπέρ κατά Α, με συγχωρείτε, η 236 δεν διαγράφει, υπήρξε έτοιμα για διαγραφή. 236 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 237 τώρα της κυρίας Λοχμπίλερ, υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε για τη 237. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Κύριε Μποργέτσιο, πρόεδρε, μπορείτε να ζητήσετε από την Ιταλική Διερμηνία να μιλά ώστε να την ακούνε. Δεν ακούμε. Τι είπατε συνάδελφε? Απεργούν Παρακαλούμε την Ιταλική καμπίνα. Μπορείτε να πείτε κάτι. Κύριε Μποργκέτσιο, ακούτε τώρα. Πολύ ωραία. Πού είμαστε? 238 Κόβατσεφ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 242 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 254 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 256 υπέρ, κατά, αποχές, 256 έλεγχος. Πέρας, εγκρίνεται. 257 σε δύο τμήματα και μάλιστα ένα εκπληκτικό ε, πεντάπτυχο. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Α, είναι free vote. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίθηκε με μεγάλη διαφορά. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μου φαίνεται ότι εγκρίνεται. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε για το πέμπτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται. 258 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 259 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε για τη 259. 259. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 260 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 265 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 266 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 267 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε για τη 267, έχετε δίκιο, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. 268 κατά Καταπίπτει. 269. σόλτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε για τη 269. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 276. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 33. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 279 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 279 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 281 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 282 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 283 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε όμως για την 283. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας εγκρίνεται. 284 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 285 υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 286 υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 287 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 288 υπέρ. Κατά. Τι έλεγχο. 287 να ελέγξουμε. Νομίζω ήταν σαφέστατο, αλλά Παρά το αποτέλεσμα, μετά το αποτέλεσμα το χθεσινό βραδινό, το καταλαβαίνω. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Με μικρή διαφορά απορρίπτεται. 288 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Ελέγχουμε Moody 288. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φτάνουμε στην 35 κιόλας. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 300 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 συμβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 309 σόλτ υπέρ Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ελέγχουμε για την 309. Ε, Πέρας. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 316 μούντι υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ξανά άρχεται η ψηφοφορία πέρας αυτής εγκρίνεται 318 έως 321 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπονται. 300... Όχι, ήταν ξεκάθαρο. 322 λοχπίλα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τώρα να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται 29 προς 28. Σχόλια εκτός μικροφώνου. 322 εγκρίθηκε, οπότε καταπίπτει. 323 για πείτε μου και 324 και 325. Οπότε φτάνουμε πάλι στην κυρία Μούντε. 326. Υπέρ, κατά. Αποχές. Έλεγχος. 326. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 30 προς 28. Πάντα μικρές οι διαφορές. 327 Λοχμπίλερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 328 Τάνοκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογικές αναφορές 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ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 και με φοβερή ταχύτητα φτάσαμε στα 16 υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. Συμβαστική 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 43 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 27 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Έλεγχος. Για βόλ. 33 υπέρ. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 34 εγκρίθηκε, 35 καταπίπτει. Συμβαστική 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην προφορική τροπολογία υπαριθμών 2 που μας υπέβαλε στην αρχή της ψηφοφορίας η κυρία Λοχπίλερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φτάνουμε επιτέλους στην ηλεκτρονική ψηφοφορία τελική για το σχέδιο που τροποποιήθηκε. Wow. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Μας λείπουν δύο συνάδελφοι. Πέρας. 29 προς 9 με 20 αποχές Συγχαρητήρια στον εισηγητή. So, we're already running 50... Ωραία. Έχουμε 15 λεπτά καθυστέρηση. Να περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία. Το σημείο 8, η κατάσταση των σχέσεων Ένωσης Κίνας. Εισηγητής ο φίλος μας ο Μπάς Μπέλντο. Μπάς θες τίποτα να πεις, όχι ωραία. Ωραία. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 104 Καστάλντο άρχεται πέρας εγκρίνεται σαφώς 110 υπέρ κατά αποχές δεκτή 115 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 14 υπέρ κατά εποχές δεκτή. Συμβαστική 15 υπέρ κατά εποχές δεκτή. Συμβαστική 16 υπέρ κατά εποχές δεκτή. 131. Μποστινάρου Λάινεν υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Να περάσουμε... Το και είναι. 133 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 134 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 139 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε Ο την Άρου Λάινεν 141 μπορεί να ιτηθούν για δεύτερη φορά σε δύο λεπτά άρχεται Έλα Κνούτ. Πέρας. Και αυτή τη φορά είναι ακόμη χειρότερα. Συμβαστική 17. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 170 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 184 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 186 Dream Team Liner Bostinaro υπέρ κατά αποχές Θα ελέγξουμε. 186 ε, ελέγχουμε λοιπόν. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται και πάλι τρει ψήφου διαφορά. 187 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά εν πάση ελέγχουμε τα 187. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Δεκτή. 27-26. 188 Λοιπόν, θα χρειαστούμε τώρα το βίντεο διαιτητή. Τι έγινε με το μηχάνημά σου. Πρέπει να προχωρήσουμε. Ε, βάση δεν χάρηκε ο κόσμος. Σάντρα. Με συγχωρείτε, δεν πρόλαβα να ψηφίσω. Άρα το ίδιο θα το αποτέλεσμα. Εγώ θα ψηφίσω υπέρ. Πρόεδρος. Ωραία. Τώρα όλοι βλέπουμε ποιος ψηφίζει και ποιος δεν ψηφίζει. Για να ηρεμήσουν όλοι να ξαναψηφίσουμε. Θα πρέπει να το έχουμε κάνει βέβαια με το, στο μάτς της Γερμανίας Μεξικού, να έχουμε ξαναπαίξει το μάτς. Λοιπόν, ξαναξεκινάμε. Ελέγχουμε την 187. Λοιπόν, ελέγχουμε την 187. Δύο δεν ψήφισαν ακόμη. Τελευταία ευκαιρία. Μην μου πείτε ότι έχει χαλάσει το μηχάνημα, η κάρτα. Πέρας. 27 υπέρ, 28 κατά. Απορρίφθηκε. Ωραία. Οπότε πάμε στην 188. Πιτέρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 195 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 197. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Οπότε φτάσαμε στην 199, έτσι δεν είναι. Καταπληκτικό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 200 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σφραστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 203 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 2.12 και 2.14 υπέρ, κατά αποχές, δεκτές. 2.13 υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. 2.20 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 2.21 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 2.22 υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.41 Καστάλντ κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Ναι, αλλά εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα. Άρα ψηφίζουμε το δεύτερο. Λοιπόν, να ελέγξουμε το δεύτερο. Άρχεται. Πέρας. Προφανέστατο. Απορρίπτεται. 2.44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.46 να ελέγξουμε. Καλώς. Επιγής ειρήνη. Ελέγχουμε τη 2.46. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.48 υπέρ. Να ελέγξουμε. Κοιτάξτε, δεν περνάνε συνήθως οι τροπολογίες του Σαφάζερ, αλλά να ελέγξουμε. 2.47. Άρχεται. Πέρας. Α, ε, καλά που το ελέγξαμε. 2.48 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 2.49 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ελέγχουμε τη 2.49 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. 2.51 υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 2.52 υπέρ. Κατά εποχές Απορρίπτεται. 2.53 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 2.55 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 2.56 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 2.57 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Η Dream Team 2.58 υπέρ. Κατά αποχές. Και πάλι χάσατε. Απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Λοιπόν, συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές. Πώς είναι, το είδατε. 29, ελέγχουμε. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή, σαφώς. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. 46 και δεν θα πω ποιοι την έχουν υποβάλει. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεκτή, δεκτή, ωραία. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 59 φωτίγα άρχεται Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Α, δεν μπορώ να ψηφίσω, λέει κάποιος. Σάντρα, ακόμη και αν είχε ψηφίσει υπέρ, θα είχαμε ισοψηφία. Δεν θα άλλαζε η κατάσταση. Ωραία και πάλι για να ρεμίσουμε. Κύριε Πρέντα, για να ηρεμήσουμε θα ξανακάνουμε την ψηφοφορία. Ωραία, θα την ξανακάνουμε. Λοιπόν, άρχεται. Δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμη. Ξυπνήστε παρακαλώ. Πέρας. Ωραία. Απορρίφθηκε. 60 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 Μπίτιχόφα υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 66 άρχεται πέρας δεκτή 67 του εισηγητή Βασπέντερ υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή 70 υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 70 άρχεται την 70 πέρας δεκτή σαφώς 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική να ελέγξουμε το 73 Συμβαστική 9 λοιπόν. Υπέρ κατά αποχές, δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 86 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 86 άρχεται πέρας Μήπως δεν λειτουργεί το μηχάνημα κανένας. Σάντρα you voted. Σάντρα ψήφισες. Ε, λυπάμαι. Λυπάμαι, αλλά δεν ζητάει κανείς τίποτα. Λυπάμαι. Λοιπόν. 88-90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποχές. Τι έγινε. Πέρασε. Λοιπόν, να το ξανακάνουμε. 88, 90 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 89, Beautyhofer, επανέρχεται, υπέρ, κατά, αποχές, υπέρ. Δεκτή δηλαδή. 91, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, σαφής νίκη δεκτή 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογικές σκέψεις 1 υπέρ κατά αποχές σαν 0-0 μου φαίνεται αυτό πρέπει να το ελέγξουμε άρχεται είναι η πρώτη τροπολογία για τις αιτιολογικές σκέψεις Κανεί δεν βλέπω να ενδιαφέρθηκε για να ψηφίσει. Διαχειρό. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 1 για τι ιδεολογικέ σκέψει πέρα. 46-2 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Την 9. Άρχεται. Σάντρα. Πέρας. Δεκτή. Το 10 υπέρ. Κατά αποχές. Κι άλλο γκολ εγκρίθηκε. 11 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε όλες αυτές τις μυστηριώδεις ε, τροπολογίες της ε, γνωμοδότησης της ΣΥΝΤΑ. Ευτυχώς, ευτυχώς. Δόξα τω Θεώ. Τώρα περνάμε στην ένβη. Όχι, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε όλες μαζί. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές συστάσεις του συγητή. Αχ, ένβη μία, ένα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ένβη δύο, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ένβη 3 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. MV4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. MV5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. NV6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. NV7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ κατά, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές ε, θα την ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Ε, βλέπετε. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεν ψηφίζουμε. 15-16 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 17 υπέρ. Κατά αποχές. Ελέγχουμε τη 17. Άρχεται. Πέρα Δεκτή. 18 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 19 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 20 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 21 υπέρ. 21 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την 21. Ένβη 21 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε την 22. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 23 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Τώρα έχουμε την αιτιολογική σκέψη α υπέρ κατά δεκτή. Ε, σκέψη β υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται, αλλά θα την ελέγξουμε. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίθηκε με μικρή διαφορά. Ένα της ΕΝΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε πραγματικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκε. Και τώρα ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε το σχέδιο δηλαδή. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά, έτσι. Τρεις ακόμα μένει να ψηφίσουν. Πού είσαστε, τελευταία ευκαιρία για να ψηφίσετε σήμερα πέρα της ψηφοφορίας και εγκρίθηκε 43 ψήφοι υπέρ, 9 κατά. Συγχαρητήρια κύριε Μπέλντερ. Διαδικαστικό, ο Μίχαηλ Γκάλερ. Ναι. Θέλω να ενημερώσω τους αδέφους πριν αποχωρήσουν για την έκθεση όσον αφορά το Ταμείο Άμυνας, όπου δεν έχουμε συμφωνήσει ΑΦΕΤ και ΙΤΡΕ για την συμμετοχή. Εμείς θέλουμε την παράγραφο 55. Και τώρα το θέμα είναι ότι οι συνάδελφοι ΙΤΡΕ τεχνικά ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα που μιλάμε έτσι, να συμφωνήσουν μαζί τους και να έχουν μια τεχνική συνάντηση. Γι' αυτό και εγώ ε, ήθελα να πω ότι μια τέτοια απόφαση πριν από, την, ε, από τους πρόεδρους των επιτροπών δεν πρέπει να γίνει. Πρέπει επίσης όρις να γίνεται η αντιμετώπιση και δεν είναι σωστό να υπάρχει τέτοια συνάντηση τεχνική. Του ζήτησαν να το καταγράψουν αυτό. Οι συνάδελφοι θα πρέπει να ξέρουν τι γίνεται πριν υπάρξει τελική απόφαση από τα αρμόδια φόρα. Αυτό είχα να πω. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Μίχαλ Γκάλερ. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, όσοι δεν ενδιαφέρονται να παραμείνουν στην συνεδρίασή μας, παρακαλώ να εγκαταλείψουν ησύχως την αίθουσα. Συνάδελφοι, είναι σοβαρό θέμα. Υπάρχουν διαφορές απόψεων ανάμεσα στην Ήτρε και την ΑΦΕΤ για τις αρμοδιότητες όσον αφορά αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Χτες υπήρξε ε, συνάντηση. Δεν βρήκαμε λύση. Ο πρόεδρος Πούσεκ και εγώ θα πρέπει να το συζητήσουμε και αν δεν βρούμε λύση θα πρέπει να υπάρξει λύση από την πρόεδρο των πρόεδρων επιτροπών. Ευχαριστώ πάντως για αυτήν την ενημέρωση. Καλή ήταν η διαμαρτυρία μας πάντως. Τώρα, συνάδελφοι. Με 45 λεπτά καθυστέρηση ερχόμαστε στις ε, εκθέσεις της Επιτροπής. Συνήθως τελειώνουμε έγκαιρα την ψηφοφορία. Αυτή τη φορά κράτησε παραπάνω, δεν ξέρω γιατί. Όταν υπάρχουν τέτοιες επίμαχες εκθέσεις και ψηφοφορίες, Ίσως θα έπρεπε να σχεδιάζουμε, να προβλέπουμε περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, είμαστε στο σημείο 9, έκθεση της Επιτροπής για τη Σερβία. Συγητής για την έκθεση αυτή είναι ένας Γερμανός συνάδελφος, David McAllister λέγεται, λέει ο πρόεδρος. Θα ε, του δώσω τον λόγο λοιπόν για να μιλήσει ως εισηγητής, εφόσον συμφωνείτε. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να είμαι σύντομος, γιατί όπως είπαμε έχουμε καθυστερήσει. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι η έκθεσή μου έχει πέντε βασικά μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι η Σερβία βρίσκεται στο δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα έκανε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, πήρε σημαντικά μέτρα τους τελευταίους 12 μήνες προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Έχει προχωρήσει όσον αφορά την ελεύθερη οικονομία, έχει οικονομική ανάπτυξη και μακροοικονομική και νομισματική σταθερότητα. Όμως η προσχώρηση, η διαδικασία προσχώρησης αποτελεί έναν μεγάλο και μακρύ δρόμο και θα επιτευχθεί μόνο εφόσον υιοθετηθούν οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις. Η προσχώρηση δεν είναι ημερομηνίε, είναι αποτελέσματα και ειλικρινά ελπίζω ότι τους επόμενους μήνες θα συνεχίσει η Σερβία την διαδρομή αυτή προκειμένου να ενταχθεί. Κράτος δικαίου. Αποτελεί στοιχείο κλειδί στις διαπραγματεύσεις. Η Σερβία προσπαθεί να έρθει πιο κοντά σε εμά ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν τα σχετικά κεφάλαια ε, τα ενταξιακά. Αλλά βέβαια πρέπει να γίνουν ε, μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου. Και ακόμα και αν το Βελιγράδι δείχνει ότι θέλει να αντιμετωπίσει πολλά από τα ζητήματα, είναι ζωτική σημασία να κάνει περισσότερες προσπάθειες για να επιτευχθεί η ανεξαρτησία και η πλήρης αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης και η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Τρίτον, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης πρέπει να διασφαλιστεί. Τα επόμενα χρόνια πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τα μέσα ενημέρωση στη χώρα. Όλοι εδώ συμφωνούμε ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωση αποτελεί βασικό στοιχείο τη δημοκρατία και μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κατάλληλη νομοθεσία, αλλά δεν φτάνει. Και μόνο αυτό πρέπει να υπάρξει και το κατάλληλο κλίμα. Τέταρτο μήνυμα. Η Σερβία συνεχίζει την ε, διαδικασία προκειμένου να έχει κανονικές σχέσεις με το Πέδιο και υπάρχει επικοδομητικός εσωτερικός διάλογος προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι δύο πλευρές, και το Πέδιο και η Σερβία, πρέπει να προχωρήσουν και να εφαρμόσουν πλήρως όλες ε, τις συμφωνίες τις οποίες έχουν καταλήξει καλή την πίστη. Η δημιουργία μιας κοινότητας σε όλους τους δήμους της Σερβίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να προχωρήσει και θα βοηθήσει και τις δύο πλευρές. Και η πέμπτη μου παρατήρηση. Είμαι πεπισμένος κοινοβουλευτικός και πιστεύω ότι για το Σερβικό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να τελέσει το ρόλο του άσκησης κριτικής προς την εκτελεστική εξουσία. Αυτό πρέπει να γίνει και με τις κατάλληλες διαδικασίες να μην υπάρχουν πια εμπόδια. Και η Πρίστινα πρέπει να αναλάβει το δικό της ρόλο δημοκρατικό σώμα στον έλεγχο της νομοθεσίας. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ βασικό η Σερβία να μην αναβάλει πλέον δράσεις ή την υλοποίηση των υποχρέωσεών της προκειμένου να ευθυγραμμίσει την ε, δικιά τη εξωτερική και πολιτική ασφάλεια προς εκείνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θέλω τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσει και θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στους ε, σκιώδεις εισηγητέ. Ο κύριο Κούκαν βέβαια πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Βεβαίως. Θα είμαι κι εγώ σύντομος. Ουσιαστικά συμφωνώ με τόσα είπατε. Θέλω να πω ότι ο κύριος Μακάλιστερ έκανε όπως πάντα πολύ καλή δουλειά. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πρόσφατα με τους Σέρβους συναδέλφους για την κατάσταση στην Σερβία ε, βάσει της κοινοβουλευτικής ε, επιτροπής ε, για την σταθερότητα και τη σύνδεση. Πρέπει να πω ότι όντως έχουν, έχει επιτευχθεί πρόοδος ανοίγουν ε, κεφάλαια ε, προενταξιακά, ήδη δύο και αναμένονται άλλα δύο για φέτος. Δείχνει η Σερβία ότι όντως βοηθάει αυτή η διαδικασία στο να γίνουν αλλαγές, κάτι το οποίο αποτελεί και παράδειγμα για την περιοχή. Εκπρόσωπος της Σερβίας είπε ότι τε θέλουν αυτή τη διαδικασία και έχουν ε, τις φιλοδοξίες αυτές που πρέπει για να πετύχουν βέβαια πρέπει να ακολουθήσουν δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Ο εισηγητής πολύ σωστά ανέφερε τους κύριους τομείς όπου πρέπει να γίνουν οι αλλαγές. Κράτος δικαίου, δικαιοσύνη, δημοκρατικοί θεσμοί, καταπολέμηση διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, ελευθερία μέσων ενημέρωσης και καλές σχέσεις γειτονίας. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τη Σερβία προς τις ψηλές αυτές προδιαγραφές και να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στις μεταρρυθμίσεις, κυρίως όσον αφορά τη δικαιοσύνη και την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του κοινοβουλευτικού έργου, που πρέπει να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση έχει να κάνει και τα, με τα μέσα ενημέρωσης και για τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Όπως είπα νωρίτερα, πρέπει να περιμένουμε περισσότερες προσπάθειες από τη σερβική κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να ευθυγραμμιστεί επίσης πιο γρήγορα στις πολιτικές της με εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβανόμαστε το λέει η σερβική κυβέρνηση, αλλά θέλουμε να δούμε μεγαλύτερη δέσμευση μια που πρόκειται και για άλλε δυνάμει στην περιοχή. Οι κανονικέ σχέσεις με το Κωσυφοπαίδιο βρίσκονται επί και καταλαβαίνω ότι θέλει ο εισηγητή μα και από την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση να πει περισσότερα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Η Σερβία βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να κάνει περισσότερα για να τηρήσει τις υποχρεώσεις της προκειμένου να ελοπιθούν οι μεταρρυθμίσεις. Προτείνω οι σερβικές αρχές να δουλέψουν περισσότερο ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνδυτοποίηση των αποτελεσμάτων από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κούκαν και ευχαριστούμε πολύ που προεδρεύσατε και τη συνάντηση αυτή της προηγούμενης εβδομάδας στο Στρασβούργο. Συναδελφοί, τώρα περνάμε στα σχόλια. Εντεκάμιση το πολύ πρέπει να σταματήσει η συζήτηση για τη Σερβία, γιατί μετά έχουμε ακόμα το Κωσυφοπέδιο και την Αλβανία. Δύο λεπτά ο καθένας, λοιπόν, παρακαλώ, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό, ο πρώτος εκ μέρους των σοσιαλιστών, ο κύριος Φλέγκενστάιν, είναι στον κατάλογό μου, αλλά δεν είναι παρόν στην αίθουσα. Καλά. Μετά. Από το ECR δεν έχει ζητήσει το λόγο. Άλντε. Ο Ιβο Βάγκλεχ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να υπογραμμίσω με τη σειρά μου ότι προετοιμάσαμε πολύ καλά την έκθεση αυτή, ο πρόεδρός μας δηλαδή, και συγχαρητήρια για αυτό, πρόεδρε. Θέλω να ανακοινώσω ότι η ομάδα μας θα υποβάλει διάφορες τροπολογίες. Αυτό γιατί η σερβική κυβέρνηση και οι αρχές γενικά πρέπει να ξέρουν ε, ότι δεν τους προσκαλούμε σε δωρεάν γεύμα, ότι πρέπει να συμμορφωθούν με τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ε, πολλοί τομείς όπου δεν συμβαίνει όμως αυτό τα μέσα ενημέρωσης, για παράδειγμα, η δικαιοσύνη, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι μερικά μόνο παραδείγματα. Έχω στοιχεία από την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών και για το 2012 από ό,τι φαίνεται υπήρξαν 81 δολοφονίες που σχετίζονται με την μαφία και μόνο 6 από αυτά έχουν διαλευκανθεί από αυτά τα εγκλήματα. Επίσης, θέλουμε να βοηθήσουμε και στη διατύπωση όσον αφορά την ευθυγράμμιση με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για παράδειγμα σε σχέση με τις υπερβολικές ενδείξεις φιλίας απέναντι στην Ρωσία. Και για τα μέσα ενημέρωση, δεν πιστεύω ότι φτάνει να λέμε ότι δεν έχει υπάρξει πρόοδος. Είναι ένα καυτό ζήτημα στη Σερβία. Και θα έπρεπε να το υπογραμμίζουμε και αυτό στις εκθέσεις μας και στις συζητήσεις μας. Ολοκληρώνοντας, Θέλω να πω ότι φυσικά και μας ενδιαφέρει η πρόοδος της Σερβίας προκειμένου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια σημαντική χώρα και ένα σημαντικό εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ιβο Βάγκλ. Ισκιώδης εκ μέρους των Πρασίνων, ο κύριο Σόλτες. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή μας που ετοίμασε το σχέδιο αυτό έκθεσης. Νομίζω ότι είναι καλά ισορροπημένη η έκθεση αυτή και αναφέρει τους διάφορους τομείς που όντως πρέπει να υπογραμμιστούν. Συμφωνώ και εγώ ότι η Σερβία βρίσκεται στο σωστό δρόμο προς την ευρωπαϊκή ένταξη, ότι έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος, έχουν ανοίξει νέα κεφάλαια. Όπως είπε και ο εισηγητής, η πρόοδος έχει προχωρήσει όσον αφορά την ελευθερία της οικονομίας, υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, σταθερότητα στη χώρα. Γίνεται καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, όμως ε, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Εξαιτίας τώρα κάποιων πληροφοριών που έχουμε από την κοινωνία των πολιτών, από μη κυβερνητικέ οργανώσει, φαίνεται να μην υπάρχει μεγάλη πρόοδο. Θα έλεγα μάλιστα ότι υπάρχει έλλειψη πρόοδου στην ελευθερία του τύπου. Και εξακολουθούν να υπάρχουν απειλέ απέναντι σε δημοσιογράφους. Συμφωνώ και εγώ με τον εισηγητή για το ότι η Σερβία θα πρέπει να επιταχύνει τους ρυθμούς υλοποίησης μεταρρυθμίσεων στο κράτος δικαίου και την ε, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Να υπάρχει διαφάνεια και οι πολίτες να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στο κράτος και στη δημοκρατία. Υπάρχει βέβαια και το θέμα των σχέσεων Σερβίας Σερβίας-Κοσυφοπεδίου. Θα το πω και αυτό. Και πραγματικά προσβλέπω στη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, Βελιγραδίου και Πρίστινα. Και αυτό έτσι ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Ελπίζω αυτή τη βδομάδα και την επόμενη βδομάδα να υπάρξει κάποια πρόοδος σε αυτό. Και τέλος, ως μέλος των Πρασίμων, θα ήθελα κάτι παραπάνω όσον αφορά το περιβάλλον. Νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση στο θέμα του περιβάλλοντος, οπότε και εμείς θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες στην έκθεση αυτή και βέβαια προσβλέπουμε και εμείς σε καλή συνεργασία με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους σκιώδης. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σόλτες. Από το Ιευθυντή ο κύριος Καστάλτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ και για την εξαιρετική σας δουλειά. Η Σερβία είναι από τις πρωταγωνίστριες ε, και τις πρωταθλήτριες μαζί με το Μαυροβούνιο στην προσπάθεια ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αξιολογήσουμε όμως τα βήματα πρόοδο που έχουν γίνει ως τώρα για την κάθε μια από τις υποψήφιε χώρες ε, προς την προσχώρηση. Πρέπει να ζητήσουμε να ισχύει αρχή more for more και less for less όμως. Από το 2014 ξεκίνησαν, άνοιξαν μάλλον 12 κεφάλαια, εκ των οποίων δύο έχουν κλείσει. Σαφής ένδειξη της δέσμευσης στον δρόμο προς την ένταξη. Να υπογραμμίσω ότι με το πακέτο διεύρυνσης που ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες η Επιτροπή ξεκίνησε η συνταγματική μεταρρύθμιση που αυτή τη στιγμή εξετάζει η Επιτροπή της Βενετίας και που αποδείχτηκε ότι είναι μια σφαιρική διαδικασία, συνολική διαδικασία που συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών. Επίση για τα θέματα τη δημόσια δίκη, τη καταπολέμηση τη διαφθορά, τη διαφάνεια, για την ε, αναθεώρηση του ποινικού κώδικα και την καταπολέμηση του εργανομένου εγκλήματο καθά και τι έρευνε και διώξει εγκλημάτων πολέμου έχουν γίνει σημαντικέ πρόοδοι. Άλλη θετική πτυχή, ένα πρόγραμμα δράση για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όπω και την κοινωνική ε, συμπερίληψη των ε, ε, μειονοτήτων των Ρωμά. Θα πρέπει να δούμε τι βήματα έχουν γίνει για την ελευθερία τη έκφραση επίση και για την άνθηση των μέσων μαζική ενημέρωση που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πολυφωνική και συμ... ένα Πολυφωνικό κόσμος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που να συμμετέχουν όλοι. Θα πρέπει να υπάρξει σταθεροποίηση και πολλές ε, πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο. Η εξομάλυνση των σχέσεων με το κοσφοπέδιο είναι σημαντική, την επανέλαβε και ο πρόεδρο Βούτσιτ στα πλαίσια του εσωτερικού διαλόγου με το κοσφοπέδιο, που θα πρέπει να οδηγήσει σε μια φάση ανάπτυξη και αναθέρμανση των σχέσεων αυτών. Ελπίζουμε να υπάρχει μια δεσμευτική συμφωνία στο θέμα αυτό και εμπιστοσύνη καθοριστική σημασία για τη σταθεροποίηση τη ευρύτερη περιοχή και προκειμένου να υπάρξει ένταξη μακροπρόθεσμα. Για τι σχέσει Σερβία και Ρωσία τώρα, όταν ζητάμε από τη Σερβική κυβέρνηση να ευθυγραμμιστεί στην εξωτερική πολιτική τη Ένωση, δεν θα πρέπει να ε, θεωρούν ότι τους ζητούμε να επιλέξουμε μεταξύ και της Ρωσίας ή προσπαθούμε να τους τριμώξουμε στη γωνία. Απλώς θέλουμε ε, ο παραδοσιακός δεσμός που έχει η χώρα αυτή με τη Ρωσία να την μετατρέψει σε μια γέφυρα για τις σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία. Να κλείσω λέγοντας για άλλη μια φορά ότι εύχομαι ότι καλύτερο για την πορεία προσχώρησης της χώρας και θα παραμείνω ένας ένθερμος υποστηρικτής της. Ευχαριστούμε τον κύριο Καστάλντο από το ΕΛΚ. Ο κύριος Ντέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας επενέσω κι εγώ για την εργασία σας. Ήταν ε, ιδιαίτερα ισορροπημένη η έκθεση, αλλά ένα σύντομο σχόλιο καταρχάς. Στο Κοινοβούλιο πάντοτε ήμασταν πολύ ένθρωποι υποστηρικτές του ανοίγματο ε, διαφόρων κεφαλαίων, παρόλο που ε, υποστηρίζαμε ότι πρέπει να βασιστούμε σε συγκεκριμένα στοιχεία για να υπάρξει πορεία ένταξη. Εδώ ανοίξαν το κεφάλαιο, το 23 συγκεκριμένα, και είδαμε ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, όμω έχει γίνει δουλειά για τι εθνοτικέ μειονότητε και τα συμβούλια του. Ε, ενώ μιλάμε τώρα, το Σερβικό Κοινοβούλιο εγκρίνει νόμους που είναι σημαντικό μέρος του προγράμματος δράσης ε, και όσων προβλέπει το κεφάλαιο 23. Γνωρίζουμε ότι τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων είναι τεράστια σημασία για την περιοχή και για όλα τα γειτονικά κράτη-μέλη. Κατά την άποψή μου λοιπόν υπάρχει βελτίωση στο κεφάλαιο 23, ε, υπάρχει πρόοδος και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν λάβει τις αποφάσεις του Συμβούλου για το άνοιγμα άλλων κεφαλαίων. Ευχαριστώ. Α, τώρα μπορώ να δώσω το λόγο στον Κνούτ Φλέκενσταν που επανήλθε. Δυόμιση λεπτά παρακαλώ για τους εκπροσώπου των ομάδων. Δεν θα τα χρειαστώ καν. Πολύ καλή έκθεση, κύριε Πρόεδρε, η δική σας. Συμφωνώ με όλα όσα αναφέρει. Είναι σαφές ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας για το κράτος δικαίου και για άλλα. Όλοι είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό. Αλλά, από την άλλη μεριά, πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει υπάρξει σαφής πρόοδος. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θέμα της σταθερότητας της περιοχής. Τώρα βέβαια, επευκαιρία, θέλω να αναφερθώ στις σχέσεις Βελιγραδίου-Πρίστινας. Όλοι το αναφέρατε. Αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην λέμε πολλά, να μην υπογράφουμε πολλά και μετά να μην εφαρμόζουμε αυτά τα οποία λέμε. Για να εφαρμοστεί κάτι δεν εναπόκειται μόνο το κάθε κείμενο στην κυβέρνηση του Βελιγραδίου, αλλά και στις αρχές της Πρίστινα. Ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ανοίξουμε την επόμενη εβδομάδα και μερικά νέα κεφάλαια. Είναι σαφής η άποψή μας από αυτού και ας δούμε τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ε, Κνούτ Φλέκενστάιν. Επόμενος ομιλητής του ΕΛΚ είναι ο Κριστιαν Ρέντα. Καταρχάς να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε για αυτή την έκθεση. που αναφέρει και τα θετικά και τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας, ε, προκλήσεις που είναι πολύ άριθμες ακόμη, όπως το είπαν ήδη οι συνάδελφοι. Για παράδειγμα, πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένα οι μεταρρυθμίσεις και αναμένουμε προόδους για το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ε, ελευθερία έκφρασης των μέσων. Όπως είπε και ο Σάλφος Ντέλη, πρέπει να γίνουν διάφορα και για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, για την εκπαίδευση, τη χρήση των γλωσσών τους και την ε, πρόσβαση στις ε, θρησκευτικέ ε, τελετές. Πρέπει η δέσμευση της Σερβίας πρέπει να είναι απόλυτη και πρέπει να τη βοηθήσει η Ένωση σε αυτή την προσπάθεια. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος της Βουλγαρικής Προεδρίας να μπορέσουμε να ανοίξουμε πάνω από δύο κεφάλαια. Ξέρω ότι οι Σέρβοι είναι ήδη προπαρασκευασμένοι για να ανοίξουν πάνω από δύο και από την πλευρά μας λοιπόν εμείς, δηλαδή το Συμβούλιο, πρέπει να έχουμε ε, ανοιχτή προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Κριστιαν. Και τώρα η κυρία Ντουμπρόφκα Ζουίτσα. Ευχαριστώ. Σε συγχαίρω για την έκθεση. Πολύ ισορροπημένη. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες. Η πρόσβαση στην Ένωση δεν είναι θέμα ημερομηνιών, αλλά γεγονότων. Αλλά έχει υπάρξει πρόοδος. Λειτουργεί η οικονομία της αγοράς, αλλά χρειάζεται περαιτέρω πρόοδος, όπως όλοι είπαμε. Πρέπει να μειώσουν την άτυπη ή γκρίζα οικονομία. Πρέπει να αναδιαρθρώσουν ε, τους νόμους για, την, ε, για, τους για τις κρατικές επιχειρήσεις και πρέπει να βελτιωθούν οι διαδικασίες και οι πρακτικές για τις δημόσιες προμήθειες. Χαιρετίζω το, την έγκριση του προγράμματος δράσης για τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων. Τονίζω το θέμα της Βόηβοντινα. Πολύ καλά όσα συμβαίνουν εκεί. Και προσβλέπω και στην εξομάλυση των σχέσεων με το Κωσυφοπαίδιο. Θα πρέπει να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Τέλος. Δεν είμαι πεπισμένη ότι η Σερβία είναι έτοιμη για να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και εξωτερικών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γι' αυτό, γιατί η Σερβία είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή. Άρα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Είναι νομίζω ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της έκθεσής σου. Ελπίζω να το κατανοήσουν. Γιατί αυτό το θέμα των σχέσεων με τη Ρωσία ξέρω ότι αλλάζει η κατάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν θέλουμε να τους έχουμε στο πλευρό μας, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ζόφκου. Τι you. Sorry, I'm, a bit um, yeah, confused. Σας συγχαίρω για την εκθεσή σας. Για το θέμα της μετανάστευσης θέλω να πω κάτι. Για το οποίο θα υποβάλω και τροπολογίες. Η Σερβία πρόσφατα κατήργησε τις ε, βίζες με το Ιράν. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις γειτονικές χώρες, ιδίως στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη όπου πηγαίνουν πάρα πολλοί πρόσφυγες. Πρέπει να τονιστεί αυτό. Πρέπει να είναι προϋπόθεση προς τη Σερβία. Πρέπει να τους συγχαρούμε για το, τη διαχείριση της ε, <coughs> μετανάστευσης, αλλά πρέπει να προσέχουν όταν καταργούν τις προξενικές θεωρήσεις με χώρες που είναι πηγή μετανάστευσης. Γιατί αυτό δημιουργεί επικίνδυνες ζωές προς γειτονικές χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο και τέλος, ο Αρνό Ντανζόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και συγχαρητήρια για την έκθεσή σας. Πολύ καλή. Εξή συντόμω. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί έναντι αυτών που ζητάμε από την κοινοβουλευτική εργασία. Ε, δίνουμε πάρα πολλέ ε, εντολέ και συνταγέ για το πώ θα λειτουργήσει το κοινοβούλιο ενό κράτου μέλου. Δεν είναι και άψογη δική μα λειτουργία. Δεύτερον, ελευθερία έκφραση και ανεξαρτησία των μέσων συμφωνούμε όλοι. Είναι ουσιώδει αρχέ του κράτου δικαίου και έχουν ιδιαίτερη σημασία. Σωστά το τονίζει η έκθεσή σα. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη Σερβία, για πολλέ χώρε τη περιοχή. Αλλά νομίζω ότι σε πολλά μα σχολεία θεωρούμε ότι η ανεξαρτησία των μέσων είναι μόνο ανεξαρτησία από την κρατική εξουσία και τις κυβερνήσεις. Η ανεξαρτησία των μέσων είναι ανεξαρτησία και από ομάδε πιέσει που δεν είναι κατά ανάγκη η κυβέρνηση. Διάφοροι ολιγάρχες, διάφορες, ε, διάφοροι όμιλοι ισχυρά, ισχυροί οικονομικά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφάνεια για την διοκτησία των μέσων, για τους μετόχους τους κτλ. Γιατί υπάρχουν ε, διάφορα μέσα που είναι ιδιαίτερα αντικυβερνητικά σε όλες αυτές τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, που έχουν απόλυτη ελευθερία έκφραση και πολλέ φορέ ε, κάνουν και κατάχρηση αυτή γιατί μα κατακρίνουν για παράδειγμα με πολύ καταχρηστικό τρόπο και το ξέρετε πολύ καλά εσεί κύριε Σιγητά και τα μέσα αυτά είναι πραγματικά ανεξάρτητα. Και τρίτον, συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Καστάλντο και την κυρία Ντουμπρόβκα για τις απαιτήσει ευθυγράμμισης με τη δική μας εξωτερική πολιτική. Όταν βλέπω την ελευθερία με την οποία ορισμένα κράτη-μέλη διαφοροποιούνται από τις κοινέ θέσει, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σχέση με τη Ρωσία, δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε υπερβολικά απαιτητικοί εναντί της Σερβίας. Είναι μια εντελώς, εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση οι σχέσεις της Ένωσης με τη Σερβία και δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε υπερβολικά απαιτητικοί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Αγνοδανζόν και τώρα η κυρία Ρουίθ Καλαβέρα από την Γενική Διεύθυνση ΝΙΑ. Ευχαριστώ κύριε Μακάλιστερ για αυτή την εξαιρετική ε, έκθεση ε, και για την αποτίμηση της δικής μας έκθεσης, για την αξιολόγηση της Σερβίας και την προοπτική ένταξής της. Αυτή η προοπτική ε, ελπίζουμε να οδηγήσει σε άνοιγμα περισσότερων κεφαλαίων μετά την τωρινή προεδρία. Ελπίζουμε ο ρυθμός διαπραγματεύσεων με τη Σερβία να μην εξαρτηθεί μόνο από το πόσο πρόοδο έχουμε επιτελέσει σε τεχνικό επίπεδο για τα διάφορα κεφάλαια, αλλά όπως έχουμε ε, πει και άλλες φορές, να εξαρτηθεί και από τη δυνατότητα της Σερβίας να προχωρήσει στο κράτος δικαίου και την εξομάλυση των σχέσεων με το κοσυφοπαίδιο. Πραγματικά είναι μια κρίσιμη συγκυρία για τις διαπραγματεύσεις με την Σερβία, επειδή έχουμε συνταγματική μεταρρύθμιση και περιμένουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα πλέον. Αναφέρατε την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, την ελευθερία των μέσων και την προστασία των εθνοτικών μειονοτήτων. Βεβαίω, ε, χαρήκαμε που στην πρόσφατη επισκέψή σα ε, τον Μάιο τα θυμήσατε όλα αυτά τα θέματα, του δώσατε έμφαση και όλος ιδιαίτερος στην λογοδοσία και τον έλεγχο της κοινοβουλευτικής ε, δραστηριότητας, κάτι που αναφέρθηκε και στην κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση. Εδώ με το Κοινοβούλιο ε, μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουμε τη διαφορά ώστε να βεβαιωθούμε ότι η διαδικασία της ένταξης βασίζεται σε θετικά στοιχεία και ότι η Σερβία όντως έχει προοδεύσει να ολοκληρώσω τονίζοντας τη σημασία της ε, ε, επικοινωνίας μας. Θα πρέπει να προβάλλουμε τα πλεονεκτήματα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο λαό της Σερβίας και ε, να παραμείνει υψηλό το φιλευρωπαϊκό φρόνημα στη Σερβία. Η κοινωνία τελικά θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο τελικός προορισμός της Σερβίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και συγχαρητήρια για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Ρουίθ Καλαμπέρα. Άλλα σχόλια από τους συναδέλφους. Ωραία, τότε να σας ευχαριστήσω για τις συνεισφορές και τις παρατηρήσεις σας. Αναμένω την εκείνη μας δουλειά για την έκθεση αυτή, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 30 Αυγούστου 11 το πρωί. Έχετε λοιπόν όλο το, όλες τις διακοπές, τη διακοπή για τις καλοκαιρινές για τη θερινή διακοπή. Ε, Στι 2 Σεπτεμβρίου, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε την πρώτη εξέταση και ψηφοφορία τον Οκτώβριο στην ΑΦΕΤ, στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Περνάμε τώρα στο σημείο 10. Ήδη προλάβαμε στο χρόνο, έχουμε 7 λεπτά καθυστέρηση μόνο, ε, έκθεση της Επιτροπής για το Κωσυφοπαίδιο. Είναι χαρά μου να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Σόλτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν ε, συνέτασα την έκθεση αυτή για το κοσυφοπαίδιο, προσπάθησα, ε, προσπαθούσα να είμαι ρεαλιστής και να εμβαθύνω στα διάφορα ζητήματα που θεώρησα ότι είναι τα πιο σημαντικά από την άποψη της πρόοδου που έχει επιτελέσει η χώρα αυτή. Βέβαια, έπρεπε να προσέξω και την έκταση του κειμένου, δεν υπάρχει περιορισμό στους χαρακτήρες, οπότε έχω κάποιες βασικές παρατηρήσεις που ελπίζω ότι θα εμπλουτίσετε και εσείς με τις τροπολογίες σας εν είδη εισαγωγής. Να πω ότι μπορούμε οπωσδήποτε να πούμε ότι το κοσυφοπαίδιο έχει κάνει θετικά βήματα ε, στο πρόσφατο παρελθόν. Πρόοδος έχει επιτελεστεί, αν και θα μπορούσε να υπάρχει και μεγαλύτερη. Υπάρχουν φυσικά πολλαπλοί λόγοι που εξηγούν αυτή την εγκατάσταση. Ε, εν μέρη τα πολιτικά κόμματα στο Κοινοβούλιο είναι χωρισμένα έτσι στην ισορροπία μεταξύ τους που είναι δύσκολο να επιτευχθεί συνένεση. Ταυτόχρονα η εσωτερική επικοινωνία είναι επίσης προβληματική σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, ένας αριθμός νόμων έχουν εγκριθεί νόμοι που πηγαίνουν στην κατεύθυνση της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ένα ακόμη στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι ε, το σημαντικό βήμα που έγινε με την κύρωση της συμφωνίας για τον καθορισμό τη χάραξη των συνόρων, ε, ιδίως ε, για το σύνδρομο το ε, Μαυροβούνιο. Σημαντικό για το καθεστώ απελευθέρωση των θεωρήσεων με το πρόστοκο σφοπέδιο. Και όλα αυτά είναι σημαντικά διότι το Κωσυφοπέδιο είναι η μόνη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων των οποίων οι πολίτες δεν μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ε, πιο συνολικά θα πρέπει να θεωρήσουν τη χώρα αυτή αξιόπιστο εταίρο εφόσον πληρούνται οι σωστές προϋποθέσεις. Θα αναλάβουμε λοιπόν και εμείς αναλόγως τις ευθύνες μας για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, εάν τηρηθούν ε, τα ξεπεφωνηθέντα. Ελπίζω ότι θα υπάρξει πολιτική βούληση, στο Συμβούλιο επίσης, και ελπίζω να προχωρήσει γρήγορα αυτή η διαδικασία. Επίση, στην έκθεση μου αναφέρομαι στο θέμα τη διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματο. Είναι ακόμα ένα πρόβλημα αυτό. Είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και στο μέλλον και νομίζω ότι έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες, θα χρειαστούν προσπάθειες για να μειωθεί ο κίνδυνος ε, να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά και γεγονότα. Επίσης για την επίδραση της πολιτικής εξουσίας στον δικαστικό κλάδο ε, και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Είναι ένα θέμα αυτό Υπάρχει όμως και ένα θέμα με την καταπολέμηση της διαφθοράς στα ανώτερα κλιμάκια. Η συνεργασία της δικαστικής εξουσίας, των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων επιβολής του νόμου είναι ε, ζωτική σημασία για το κοσυφοπαίδιο. Ελπίζουμε ότι αυτή η μορφή συνεργασίας θα συνεχιστεί και ότι θα διαλευκανθεί πολύ σύντομα ο πρόσφατος φόνος. Επίσης, πιστεύουμε ότι καλό είναι να αναφερθεί κάτι που εν μέρει ανέφερε και η έκθεση ε, για την Σερβία. Θέλουμε εξομάλυνση των σχέσεων Βελιγραδίου-Πρίστινας και θέλουμε ο διάλογος να ε, συνεχιστεί, να ξαναρχίσει μάλλον όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό θα μας φέρει πιο κοντά στον απότερο στόχο μας, που είναι και για τις δύο αυτές χώρες, για τις δύο αυτές πλευρές, να τηρήσουν τις υποχρεώσεις του διαλόγου και να γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα. Είναι σημαντικό για το διάλογο αυτό να οργανωθεί σε συνθήκες διαφάνειας. Γιατί, διότι είναι δίκαιο και σωστό να παραμένει να τηρείται ενήμερο το Κωσοβάρικο Κοινοβούλιο ώστε να μπορούν να εγκρίνουν ή να προτείνουν περαιτέρω βήματα. Ολοκληρώνοντας, να τονίσω ένα θέμα που δεν είναι άνευ σημασία. Το θέμα του περιβάλλοντος. Στην φετινή ετήσια έκθεση δίνεται κάποια έμφαση και στο θέμα αυτό. Γίνεται λόγος για την ποιότητα της ε, ε ατμόσφαιρας, του ατμοσφαιρικού αέρα στην Πρίστινα, Αυτό επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων στην Πρίστινα και είναι αποτέλεσμα της δραστηριότητας του ενεργειακού τομέα στο κοσφοπέδιο. η παραγωγή ενέργειας προκαλεί, είναι μεγαλύτερη επικυρύπανση στην περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. το πρόγραμμα για την ενέργεια και για τη χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργεια είναι ζωτική σημασία για την ε, βελτίωση του βιωτικού επίπεδου στο δοσφοπέδιο. Εάν λοιπόν γίνουν τα απαραίτητα βήματα, είμαι βέβαιο ότι σε συνεργασία με του κλάδου εισηγητέ θα καταφέρουμε να ε, βελτιώσουμε το κείμενο με τι κατάλληλε τροπολογίε και να, να καταλήξουμε σε μια ε, καλή έκθεση. Thank you, Igor Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σόλτες για την παρουσίασή σας. ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας, ο κ. Σπίτσουλ, αλλά δεν είναι εδώ βλέπω. Οπότε θα δώσω το λόγο στους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Πρέντα, πρώτα απ' όλα, από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Σόλτες για την παρουσίαση αυτή της έκθεσής του. Με εκπλήσει κάπως που βλέπω ότι σε αυτή την πρώτη εκδοχή τουλάχιστον δεν αναφέρεται τίποτα για το ότι πέντε χώρες μέλη δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσυφοπαίδιο. Είναι πέντε στις 28 μεν, αλλά είναι μία θέση Είναι μια πρακτική που ήθιστε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αναγνώριση κρατών. Έπειτα με εκπλήσει το γεγονός ότι δεν γίνεται μνήα στην χρήση, δυστυχώς στην ευρεία των δακρυγόνων. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Πριστίνα γι' αυτό. Έχει κάποια ευθύνη το Κοινοβούλιο στις πρακτικές, τις πολιτικές που είναι αποδεκτές ή όχι. Έπειτα για τον ε, διάλογο. Πριστίνα Βελιγράδη. Εννοείται ότι περιμένουμε πολλά από την υλοποίηση των συμφωνιών. Ξεκινώντας από εκείνη που έχει να κάνει με την συμμετοχή των Σερβικών Δήμων. Ελπίζω ο διάλογος που θα ξαναξεκινήσει στα τέλη της εβδομάδας θα ξεμπλοκάρει την κατάσταση. Πρέπει να προχωρήσουμε, να έχουμε θετικούς στόχους αυτό το διάλογο Πριστίνα Βελιγραδίου. Είναι κάτι προς όφελος όλων των χωρών, είτε αναγνωρίζουν είτε όχι το πεδίο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε, Κρίστιαν Πρέντα. Ο κύριος Παντζέρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ε, θεωρώ ότι το κοσυφοπαίδιο είναι αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, την οποία πρέπει να προωθήσουμε. Όμως το κοσφοπέδιο είναι κάπω και ο θερμοστάτης, μάλλον το θερμόμετρο που δείχνει πώς προχωρά ε, θετικά ή αρνητικά, η υλοποίηση όλη αυτή τη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια. Παρατηρήσεις εκτός μικροφώνου. Η γερμανική διερμηνία. Ξαναρχίζω από την αρχή. Έλεγα ότι το Κωσυφοπαίδιο είναι ένα απόσπαστο τμήμα της στρατηγικής για τα Δυτικά Βαλκάνια. Όμως, ταυτόχρονα είναι και ένα ε, θερμόμετρο, ένας δείκτης που δείχνει πώς προχωράει η στρατηγική αυτή από την σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μιλώντας προηγουμένως για τη Σερβία, είπαμε πρέπει να επιλέξουμε, ότι θα πρέπει μάλλον να επιλέξουμε μεταξύ ε, μιας προσπάθειας διεύρυνσης των σχέσεών μας, αλλά δεν πρέπει να μπλέκουμε δύο πράγματα. Ε, από τη μια να εντείνουμε εμεί τι σχέσει μα με τι περιοχέ αυτέ, για την άλλη να υπάρχουν έξωθεν επιρροέ στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, εκτό Ευρώπη. Ε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αναγνώριση από πέντε χώρε εδώ, πράγμα που δεν μου φαίνεται ότι είναι καλή προπόθεση για να ξεκινήσει ανεμπόδιστη όλη η διαδικασία ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων. Ωστόσο, επί της ουσίας, να πω ότι υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα στο κοσυφοπαίδιο, ο πολιτικός κατακαιρματισμός που έχει επηρεάσει το ρόλο και τη λειτουργία της Εθνοσυνέλευσης. Έχει επηρεάσει και τη δράση της κυβέρνησης και την αποτελεσματικότητά της. Είναι απαράδεκτες ε, οι δράσεις κάποιων βουλευτών, ακόμη και χρήση δακρυγόνων, ε, δεν βλέπω να είναι κάτι που μπορούμε να παραβλέψουμε ούτε και μπορεί να ε, τα μεταξύ των επίσημων ε, δραστηριοτήτων ενός κοινοβουλίου. Ε, πάντως, είναι καλή η κίνηση να κυρωθεί η συμφωνία για την χάραξη συνόρου με το Κωσυφοπαίδιο, με το Μαυροβούνιο και η προσπάθεια για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και της ε, διαφθοράς είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχιστεί και με αμύωτη ε, ένταση. Οι αρχές θα πρέπει να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο με εγκρίνοντα του απαραίτητου νόμου που θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το κοινοτικό κεκτημένο και το διεθνέ δίκαιο. Υπάρχει κι άλλο ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, εδώ υπάρχει νομικό πλαίσιο που είναι στο ύψο των ευρωπαϊκών προτύπων, ωστόσο υπάρχει και το πρόβλημα της τήρησης και της υλοποίησης των προτύπων αυτών. Αυτό δεν είναι αρκετά προχωρημένο. Το ίδιο και με την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθεροτυπία. Ως προς την εξομάνιση των σχέσεων με τη Σερβία, το κοσυφοπέδιο θα πρέπει να ε, συμμετάσχει στο σχετικό διάλογο με, ε, καταβάλλοντας τις ανάλογες προσπάθειες και να προσθέσω ότι όπως είπαμε και για τη Σερβία, το θέμα της Σερβίας είναι στενά συνδεδεμένο με το θέμα του κοσφοπεδίου. Τα δύο αυτά ε, συμβαδίζουν. Δεν μπορούμε να δούμε το ένα ανεξαρτήτως του άλλου. Δεν μπορούμε να ε, δώσουμε την ε, πρώτη θέση στη Σερβία, ας πούμε, ξεχνώντας το κοσφοπέδιο κάπου στο φόντο πίσω. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παντζέρη. Συνάδελφοι, να σας ενημερώσω ότι έχουμε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά την ημερησία διάταξη. Θα μπορούσαμε λοιπόν αύριο το πρωί να προσθέσουμε ένα σημείο στην ε, Ευρωπαϊκή, στην ε, ημερήσια διάταξη, μετά το σημείο 18 δηλαδή, ε, μετά από τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ να έχουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σήμερα δεν μπορεί να έρθει κανείς, αύριο μπορεί. Δηλαδή τι ώρα περίπου θα είναι αυτό, ξέρουμε. Γύρω στις 10 και μισή. Εντάξει. Ίσως η γραμματεία θα μπορούσε να ενημερώσει τους συναδέρφους γι' αυτό. Εντάξει, θα σας θέλει η πληροφορία. Καλώς, ωραία, ευχαριστώ πολύ. Οι ομιλητές τώρα για την έκθεση όσον αφορά το κοσίφο πέδιο εκ μέρους του Άλντε, ο κύριος Βάγκλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Θα ήθελα αντί για μένα να μιλήσει συνάδελφος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, λέει η κυρία Βάτμανς, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτή την καλή έκθεση. Ε, για μας το All Day η έκθεση αυτή, το σχέδιο έκθεσης αποτελεί πάρα πολύ καλή βάση Υπάρχουν διάφορα σημεία και πραγματικότητε που θα ήθελα να αναφέρω. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, ε, την ενδοικογενειακή βία, την συμμετοχή στις εκλογές, τη συμμετοχή των γυναικών γενικά. Και πιστεύω ότι όσον αφορά το ULEX, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά την εντολή. Εκπαίδευση. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία σε προσπάθειες κατά των διακρίσεων. Ε, υγεία. Και εδώ θα έπρεπε να αναφέρουμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ποιότητα των φαρμάκων και όσον αφορά την οικονομία θα ήθελα να υπογραμμίσουμε περισσότερο πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε τις ατυχείς εξελίξεις που έχουμε όσον αφορά την εθνικιστική και ακραία ρητορική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βοηθήσει στη συμφιλίωση ε, βοηθώντας ε, τις ε, διάφορες κοινότητες. Επίσης, το κοσυβοπαίδιο κάνει πρόοδο ας πούμε όσον αφορά την ε, δίκηση και την ισότητα ή την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, αγαθών ε, και των ατόμων ή την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση πάντως. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βάτμαντς. Επόμενος, από τους μη εγγεγραμμένους, ο κύριος Επιτίδιος παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε. Η έκθεση για την πρόοδο της εντάξεως του Κωσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφής και αναφέρει με ακρίβεια τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν και τα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν ούτως ώστε να ενταχθεί η χώρα αυτή κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι η ένταξη μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να γίνεται με βάση πολιτική σκοπιμότητα, αλλά με τη βάση της ανάγκης αλλά και τη πρόοδου που παρουσιάζει αυτή η χώρα. Παραδείγματο χάρη, το Κωσυβοπαίδιο είναι μια χώρα η οποία, εάν ενταχθεί, θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχά, είναι μια χώρα η οποία προέκυψε από την αφαίρεση ενός τμήματο από τη Σερβία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το Κωσυφοπέδιο είναι το λίκνο του σερβικού πολιτισμού. Άρα λοιπόν υπάρχουν προβλήματα ούτω ώστε να ευοδοθούν οι συνομιλίε που γίνονται με το Βελιγράδι. Απ' την άλλη πλευρά, αναφέρθηκε ότι δεν, δεν έχει αναγνωριστεί το κοσυφοπαίδιο από κάποιε χώρε. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό. Διότι ο τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε δημιουργεί και υπάρχει κίνδυνο να δημιουργήσει τετελεσμένα και για άλλε χώρε. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε το τι πρέπει να ζητηθεί να κάνει το κοσυφοπαίδιο, ούτω ώστε να μπορέσει να ενταχθεί ομαλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να μην δημιουργηθούν και στο μέλλον προβλήματα, διότι ήδη το Κωσυφοπαίδιο θέλει να κάνει μια συνομοσπονδία με την Αλβανία. Αυτό θα δημιουργήσει γενικότερα προβλήματα στην περιοχή, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η Αλβανία έχει επεκτατικές ε, βλέψεις προ τι γειτονικές χώρε. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να γίνει με βήματα σταθερά και προσεκτικά η ένταξη του πεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος Ζούτσα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία κλειδί. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σόλτες για την πρώτη αυτή έκθεση. Δύο στοιχεία κλειδί υπάρχουν εδώ όσον αφορά το κοσυφοπέδιο. Το πρώτο είναι ότι πέντε χώρες μέλη δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσυφοπέδιο, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και ένα άλλο είναι ότι υπάρχουν, υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην προσχώρηση της Σερβίας και την προσχώρηση του κοσυφοπεδίου. Είναι συνδεδεμένα αυτά τα δύο. Αν δεν υπάρξει εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Αυτά τα δύο λοιπόν στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Και αυτό το οποίο για μένα λείπει από την έκθεση είναι το εξή. Μιλάτε για γεφύρωση. Ε, μιλάτε για τους δήμους στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο. Δεν υπάρχουν όμως αυτά τα στοιχεία μέσα στην έκθεση και θα έπρεπε. Ε, χαίρομαι βέβαια για την πρόοδο όσον αφορά τη χάραξη συνόρων με το Μαυροβούνιο. Αν δεν υπάρξει όμως περισσότερη ελευθέρωση δεν θα βοηθήσει τίποτα. Οπότε ευχαριστώ για αυτά που λέτε όσον αφορά την κατάργηση της θεώρησης. Νομίζω ότι θα υπάρξουν τροπολογίες πράγματι μέσα στους επόμενους μήνες προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Φλενκστάιν. Για την ομάδα μου τα είπε σχεδόν όλο ο κύριο Παντσέρη. Να αναφερθώ λίγο σαφέστερα <clears throat> από ότι οι προηγούμενοι ομιλητές σε ένα σημείο. Και για τα άλλα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων ισχύει ότι πρέπει να παραμείνουμε αξιόπιστοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν έναντι του κοσυφοπεδίου θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι δηλαδή, εάν εκεί καλούμε για να γίνουν μεταρρυθμίσεις και μετά πραγματοποιούνται, τότε πρέπει και εμείς να παραμείνουμε αξιόπιστοι. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε το εξή. Πρέπει να θέσουμε σαφώς τις προϋποθέσεις και εφόσον προχωρήσουν τα πράγματα, θα πρέπει να υπάρξει φιλελευθεροποίηση για τις βίζες. Γιατί είναι η μόνη χώρα της περιοχής ε, της οποίας οι κάτοικοι δεν μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα. Και κάθε φορά που μας λένε τι θα γίνει με την κατάργηση, τους λέμε «Ε, κάτι ακόμη πρέπει να κάνετε. Τώρα πρέπει να λύσετε το πρόβλημα των συνόρων με το Μαυρογένιο. Και το έλυσαν. Άρα δεν έχουμε κανένα λόγο να μην στείλει φέτος το καλοκαίρι ένα σαφές μήνυμα το Συμβούλιο ότι θα υπάρξει κατάργηση των, ε, στις βίζες. Ευχαριστώ κύριε Φλέκενστάιν. Τρεις ακόμη ομιλητές. Βάγκελ, Κούγκαν και ο κ. Μποστινάρο. Εντάξει, θέλει κανεί άλλο το λόγο. Ωραία, Βάγκελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεση. Βάλτε τα ακουστικά σας για να με καταλάβετε. Η συνάδελφος, η κυρία Βάτμαν, υπογράμμισε τα πιο σημαντικά ζητήματα όσον αφορά την ομάδα μας. Πρόκειται για την οικονομική σταθεροποίηση του κοσυφοπεδίου, για να μπορεί να είναι τέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ πριν από μένα είπαν ότι η σχέση ανάμεσα στη Σερβία και το κοσυφοπέδιο είναι πολύ σημαντική και ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο είναι σημαντικός. Ότι θα επηρεάσει τις ευρωπαϊκές προοπτικές τόσο του Κωσυφοπεδίου όσο και της Σερβίας. Σήμερα όμως μιλάμε για το Κωσυφοπέδιο. Συνεπώς, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το τμήμα της τέως Ιουγκοσλαβίας να παραμείνει η ευρωπαϊκή προοπτική. Η έκθεση περιλαμβάνει διάφορα ευρήματα, τα οποία είναι δείχνουν ότι υπάρχει μια σχετική και αντικειμενική πρόοδος, παρόλο που αυτή δεν είναι πάντα αρκετή. Μην ξεχνάμε όμως ότι το Κωσυφοπαίδιο ήταν ακριβώς η λιγότερο ανεπτυγμένη περιοχή της Γιουγκοσλαβίας, της οποίας ήταν μέρος πριν. Συνεπώς αυτό μην το ξεχνάμε και πρέπει να δείξουμε σεβασμό απέναντι στο Κωσυφοπαίδιο. Αξίζει σεβασμό και από το Βελιγράδι. Και αυτό πρέπει να φανεί στις σχέσεις Πρίστινα και Βελιγραδίου. Τώρα, οι σχέσεις και ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ακούμε ότι αυτό συνήθως γίνεται στην πλευρά του κοσφοπεδίου. Ναι. Όσοι όμως είναι σημαντικοί παράγοντες σε αυτές τις συναντήσεις είναι συνήθως από την Σερβία. Ε, όταν δημιουργούνται προβλήματα, ακούμε ότι γίνονται συνήθω στο Πέδιο. Ναι, αλλά αυτοί που τα δημιουργούν είναι συνήθω από τη Σερβία. Τέλο, θέλω να πω κάτι ακόμα. Δεν καταλαβαίνω την Ισπανία και τις επιφυλάξεις που έχει απέναντι στις ευρωπαϊκές προοπτικές του Πεδίου. Προσπαθούν να παρουσιάσουν ε, και να κάνουν συγκρίσει ανάμεσα στο Κωσυφοπαίδιο και τόσα συμβαίνουν στο εσωτερικό τη ισπανία με την Καταλωνία και τη χώρα των Βάσκων. Το Κωσυφοπαίδιο είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θα πρέπει να επηρεάζει η κατάσταση αυτή τη ισπανία στις ευρωπαϊκές προοπτικέ του Κωσυφοπαιδίου. Ευχαριστούμε ο κύριο Κούκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω να κάνω μερικέ παρατηρήσει. Ευχαριστώ τον Ιγκόρ Σόλτε για την ε, καλή του έκθεση. Υπογραμμίζει την ε, ταραχώδη εποχή από την οποία πέρασε το Πέδιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά εγώ θα περίμενα μεγαλύτερη πρόοδο. Ε, περισσότερη πολιτική ηγεσία από πλευρά του κοσυφοπεδίου. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε να υπάρχει μια πραγματική ειλικρινής δέσμευση, κυρίως στο θέμα του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι πολιτικοί ηγέτες επίσης θα πρέπει να δείξουν τη δέσμευση υπέρ του κοινοβουλευτισμού. Οι συναντήσεις που έχουμε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιπροσωπεία του Κωσυφοπεδίου είναι κρίμα να μην μπορούν να καταλήγουν σε κοινή δήλωση. Από την άλλη, θέλω να συγχαρώ το Κωσυφοπεδίο για τις επικοδομητικές διμερείς επιτέλους σχέσεις όσον αφορά τη χάραξη συνόρων με το Μαυροβούνιο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ότι ευθυγραμμίζονται και με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Ε, το είπε νομίζω ο κύριος Φλέκενστάιν. Ε, πρέπει να υπάρχει μια αντικειμενική αντιμετώπιση των δύο πλευρών. Ειλικρινής διάλογος. Θα πρέπει να υπάρχει ίδια και από πλευρά Σερβία και από πλευρά του Κωσυφοπεδίου. Δηλαδή, εμεί στι εκθέσει μα να έχουμε την ίδια διατύπωση. Γιατί οι Σέρβοι λένε ότι τα βάζουμε κυρίω με αυτού, το Κωσυφοπέδιο λέει ότι τα βάζουμε κυρίω με εκείνου. Οπότε αυτό πρέπει να λυθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση το κοσιφοπεδίο να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αυτό. Τέλος, διαπίστωσα ότι οι κύριοι ομιλητής για το μέλλον του κοσυφοπεδίου χρησιμοποιούν τη λέξη ελπίδα. Η ελπίδα δεν φτάνει. Πρέπει να υπάρχουν πιο απτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Κούκαν, ο Βίκτορ Ποστινάρο τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε, έχω δύο παρατηρήσεις. Να αρχίσω πρώτα από αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, Κούκαν. Μίλησε για ελπίδα. Ε, ναι, ας πάμε όλοι μα καλύτερα, πρόκειται μόνο για ελπίδα και πίστη. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο πλευρές, αλλά και για μας, είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να υποκαταστήσει τη συμφιλίωση ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Πρίστινα. Τίποτα. Αγγίση γι' αυτό. Καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να γνωρίσει αυτό το παράγοντα που εμποδίζει τις δικές τους συνομιλίες και τις επιπτώσεις που αυτές ε, έχουν στο μέλλον τους για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και αξίζει να το υπογραμμίσουμε περισσότερο όσον αφορά την ε, πρόοδο δηλαδή των διαπραγματεύσεων. Δεύτερον, στρατηγικά δεν μπορούμε να δούμε τα Δυτικά Βαλκάνια να εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει μια τρύπα. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε αυτή την εισίδα απομονωμένη και να την ε, ξεχωρίσουμε από ένα σύνολο που θα ενταχθεί κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο παράγοντας χρόνος ε, παίζει σημαντικό ρόλο για ολόκληρη την περιοχή αν δεν υπάρξει πρόοδος στην προσέγγιση μας απέναντι στο κοσυφοπαίδιο. Και τέλος, θέλω να απαντήσω στον συνάδελφο Βόγκαλ οι πέντε χώρες που δεν αναγνωρίζουν. Συνάδελφοι, δεν είναι τόσο και το Κωσυφοπαίδιο. ίσως να μην έχει να κάνει με τις σχέσεις μας με το Κωσυφοπαίδιο. Οι λόγοι μη αναγνώριση του Κωσυφοπαίδιου έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο οι πέντε αυτές χώρες βλέπουν το θέμα του διεθνούς δικαίου και τις διατάξεις περί αυτοδιάθεσης και απόσχησης. Γι' αυτό εγώ θέλω να κάνω έκκληση στην Επιτροπή μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, να σκεφτούν τι διατάξεις, τι εγγυήσει μπορούμε να προσφέρουμε στις πέντε χώρες που δεν αναγνωρίζουν, ώστε να βάλουν στην πάντα τις επιφυλάξεις τους. Γιατί επαναλαμβάνω, η χώρα μου, η Ρουμανία, δεν έχει καμία τίποτα κοινό με το κοσυφοπέδιο, δεν έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας, διενέξεις, αντιπαραθέσεις. Κι όμως, πρόσφατα, ο πρόεδρός μας πρότεινε να βοηθήσουμε τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ από πλευράς της Πρίστινα είχαμε αρνητικές αντιδράσεις. Είναι σημαντικό όμως να κάνουμε το ερώτημα, γιατί όχι και να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα που μπορεί να διευκολύνει τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρο. Ρουίθ Καλαβέρα τώρα από την Γενική Διεύθυνση ΝΙΕΡ. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σόλτες για αυτήν την ε, πολύ καλή έκθεση, το σχέδιο έκθεσης που λαμβάνει υπόψη τα με ευρήματα και τα δικά μας. Ήμουνα πριν από δύο εβδομάδες στο κοσυφοπέδιο και η υποδοχή ήταν πολύ καλή. Συμφωνώ ότι βλέπουμε θετικές εξελίξεις στο κοσυφοπέδιο. υπάρχει ένα θετικό κλίμα και το πιο σημαντικό η επικύρωση της συμφωνίας με το Μαυροβούνιο για τα σύνορα. Τώρα ο βηματισμός για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ήταν ε, χαμηλός. Όντως υπάρχει και πόλωση στην Πρίστινα μετά τις εκλογές. Πάντως πρέπει να θαρρύνουμε το κοσυφοπέδιο ώστε να συνεχίσει τις ε, μεταρρυθμίσεις του προς την κατεύθυνση της Ευρώπης. Για μας πρέπει οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις να σταθεροποιηθούν, να προχωρήσουν και να μην υπάρχει τίποτα που θα υπονομεύσει την οικονομική σταθερότητα μεσοπρόθεσμα. Αυτό το κοίτανε και οι δύο πλευρές. Οι μεταρρυθμίσεις στη δίκηση είναι σημαντικές και βέβαια και όσον αφορά το κράτος δικαίου. Τώρα, για τα σχόλια που κάνατε για το περιβάλλον, η ΝΙΕΡ δίνει μεγάλη σημασία στην ευημερία των κατοίκων του Κοσφοπεδίου, γι' αυτό και συζητάμε με τις αρχές και λέμε ότι πρέπει να υπάρχει πράγματι μια ενεργειακή πολιτική που να περιλαμβάνει τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας και να περιλαμβάνονται στο ενεργειακό μείγμα. Και είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να τους βοηθήσουμε. Πολύ χαίρομαι που έχουμε 10 εκατομμύρια για την ενεργειακή επάρκεια του Κωσυφοπεδίου, ώστε να βοηθηθεί η κατάσταση σε όλα τα δημόσια κτίρια, να υπάρχει επαρκής ενεργειακή απόδοση, να μην χάνεται ενέργεια χωρίς λόγο. Συμφωνώ με τα σχόλια της κυρίας Βάουτμαν επίσης για το πόσο σημαντικό είναι το θέμα της νοοτροπίας προκειμένου να επιτευχθεί η συμφιλίωση και η οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό και ζητώ ζητήσαμε από το Συμβούλιο Συνεργασίας να έχει ένα πραγματικό πιλωτικό πρόγραμμα προενταξιακά προκειμένου να δημιουργηθεί μια προσφορά ε, όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Ε, κάτι το οποίο θα ευνοήσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να προωθήσουμε όχι μόνο τα ταξίδια του κόσμου ώστε να υπάρξει καλύτερη επαφή στην περιοχή μεταξύ όλων, αλλά και οι δικοί μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι πολίτες να πάνε περισσότερο. Τώρα, κατά τα άλλα, ξέρετε πάρα πολύ καλά και είναι προτεραιότητά μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην διερευνητική αποστολή που πήγαμε, ετοιμάζουμε αξιολόγηση ε, της κατάστασης όσον αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες του Κωσυφοπεδίου. Ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να έχουμε την αξιολόγηση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ρουίθ Καλαβέρα. Τώρα, Ίγκο Σόλτες, για να συνοψίσετε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, τους κοιόδης εισηγητές όλους για τα σχόλια τους. Απλώς να πω ότι επειδή ήταν ε, συγκεκριμένα τα όρια στους χαρακτήρες για, για το κείμενο αυτό, δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν όλα. Πιστεύω όμως ότι θα υπάρξουν επικοδομητικές τροπολογίες που θα βελτιώσουν το περιεχόμενο. Απλώς μια κουβέντα στο τέλος. Νομίζω ο κύριος Φλέκενστάιν είπε κάτι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να παραμένει εξόπιστος εταίρος στο διάλογο αυτό. Διότι έτσι θα ε, εκπλώσουμε καλύτερα και τις υποχρεώσεις μας. Είναι καλή στιγμή το κοσφοπέδιο να υποφεληθεί από την απελευθέρωση των καθεστώτων θεωρήσεων. Ευχαριστούμε κύριε Σολτές. Κάνατε μια κέρια παρατήρηση. Μεγάλη πρόκληση για όλους τους ηγετές αυτές τις εκθέσεις είναι ότι έχουμε περιορισμένο αριθμό χαρακτήρων ε, για αυτές τις εκθέσεις. Οπότε θέλοντας κανείς να εκφράσει όλε τι παρατηρήσεις μπορεί να πει πάρα πολλά. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κανένα όριο ε, στην έκταση των κειμένων της. Ε, δεν υπάρχει όριο. 100, 200, 500 σελίδε, άμα θέλετε. Γι' αυτό λοιπόν κάθε φορά ε, δεχόμαστε επικρίσει ότι δεν έχουμε μπει στι λεπτομέρειε του κάθε προβλήματο και φαινομένου. Ε, συνάδελφοι, ε, το πρόγραμμα για την έκθεση προοικοσφοπεδίου είναι ακριβώ το ίδιο με αυτό τη Σερβία, 30 Αυγούστου, 11 το πρωί για την των ε, επόμενο σημείο, και μάλλον θα ολοκληρώσουμε στις 12.30, έκθεση ε, για την Αλβανία και χωρίς καθυστερήσεις δίνω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Φλέκενστάιν. Αγαπητοί συνάδελφοι, την Κυριακή θα έχουμε την ε, τέταρτη επέτειο από την αναγνώριση της Αλβανίας ως επισήμου υποψηφίου. Έχουν περάσει λοιπόν τέσσερα χρόνια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη. Και ως εισηγητής χαιρετίζω αυτή τη σαφή δήλωση προθέσεων και στηρίζω αυτήν την ε, σύσταση και για λόγους προσωπικής ε, αντίληψης. Και δεν είναι κάτι που το στηρίζει μόνο η ομάδα μου, αλλά και πολλοί συνάδελφοι από το ΕΛΚ, την ΑΛΔΕ, από τους Πρασίνους. Πρώτη φορά το διαπίστωσα αυτό. Νομίζω ότι και στις προηγούμενες συζητήσεις αποδείξαμε ότι αυτό δεν είναι θέμα κομματικών σκοπιμοτήτων. Καλό θα ήταν αυτό να το έχουν καταλάβει και όλοι στην ε, Αλβανία Χαίρομαι που υπάρχει ευρεία τέτοια συνένεση γι' αυτό. Αξίζει η Αλβανία να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αν και όλοι καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι πολλά δεν είναι όπως θα έπρεπε, όπως θα το ήθελε και η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο και εμείς. Πρώτον, η Αλβανία ξεχωρίζει από τις άλλες χώρες της περιοχής, διότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σταθερές πρόοδοι για την ε, υλοποίηση των ε, μεταρρυθμίσεων που ζητήσαμε και ιδιαίτερα για τις προτεραιότητες κλειδί. Και δεύτερον, η Αλβανία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εφαρμόσει μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση στο τομέα της δικαιοσύνης που είχε προτείνει η Κομισιόν το, από το 2014 και το είχε ε, θέσει ως προϋπόθεση. Η διαδικασία μεταρρύθμισης ε, της δικαιοσύνης είναι ήδη εν πλήρη εξελίξη και έχουμε ήδη όχι μόνο τα πρώτα αποτελέσματα, αλλά έχει και ήδη ένα πολύ θετικό αντίκτυπο αποτροπής για τους εγκληματίες. Είναι λοιπόν καλό σημείο για το μέλλον. Για τη δημόσια διοίκηση. Έχει υπάρξει ήδη σε μεγάλο βαθμό μεταρρύθμιση. Οι επιτυχίες τώρα βέβαια πρέπει να μεταφραστούν και σε τοπικό επίπεδο. Ίσως θα διαρωτάστε γιατί αναφέρομαι τόσο συγκεκριμένα στην μεταρρύθμιση δικαιοσύνη. Το κάνω αυτό γιατί η πολιτική βούληση για μια τόσο σημαντική και μακρόπνοη μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη και καταδεικνύει την ευρωπαϊκή φιλοδοξία όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά συνολικά του Κοινοβουλίου δηλαδή συμπεριλαμβανομένης και της ε, αντιπολίτευση τότε που αποφασίστηκε. Ομόφωνα το Κοινοβούλιο λοιπόν προωθεί αυτήν την ε, μεταρρύθμιση. Και έτσι τίθεται ένα θαυμάσιο πρότυπο και για άλλες υποψήφιε χώρε. Άρα επηρεάζει τη συνολική μας στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και τρίτον, αυτή η μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνη έχει και επιπτώσεις θετικές και σε άλλες ε, κύριες προτεραιότητε. Επηρεάζει Ξέρουμε ότι πολλά πρέπει να γίνουν για καταπολέμηση διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Αλλά χωρίς μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη αυτοί, αυτές οι προσπάθειες δεν θα καρποφορήσουν. Στην έκθεσή μου ανέφερα και τα σημεία όπου γίνεται πρόοδος και για τα σημεία που πρέπει να υπάρξει ε, γενικότερη πρόοδος. Εδώ ε, βεβαίω πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης. Αν μια επιχείρηση θέλει να επενδύσει στην Αλβανία, πρέπει να υπάρχει αναγκαία νομική βάση για να υπάρχει εμπιστοσύνη. Και εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Επειδή έχω την ευκαιρία να τονίσω, επειδή επίκειται τη συνεδρίαση του Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα, οι μεγάλες ομάδες του σώματός μας έχουν εκφραστεί σαφώς. Η Κομισιόν επίσης. Οπότε, παρακαλούμε το Συμβούλιο να μην ξαναμπλέξει τα πράγματα τώρα με διάφορες προφάσεις, αναμαρτίες και καλλιλογικά στοιχεία. Να πει ότι πρέπει να υπάρξει έναρξη των διαπραγματεύσεων για την Αλβανία και για την Μακεδονία και ένα σαφές μήνυμα προς το κοσφοπέδιο πρέπει να είναι η απελευθέρωση των θεωρήσεων και το άνοιγμα κάποιων κεφαλαίων για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Φλέκενστάιν, για τη σύντομη παρουσίαση τη έκθεση για την Αλβανία. Λοιπόν, ποιοι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, θέλουν το λόγο. Οι συνάδελφοι Κούκα, Μποστινάρου, Σόλτε, Χατζηγεωργίου, Σακοράφα, επιτίδιος. Αυτοί. Έξι ομιλητέ. Λοιπόν, προτείνω ο καθένας ε, δύο λεπτά παρακαλώ. Κούκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Κνούτ Φλέκενστάιν που εκπώνησε αυτήν την έκθεση με σωστά και ε, ισορροπημένα μηνύματα για την κατάσταση των πραγμάτων στην Αλβανία. Θα το πω ξεκάθαρα να δώσουμε ημερομηνία για την άνοιξη διαπραγματεύσεων ε, στην Αλβανία, διότι έχει σημειώσει πρόοδο στην διαδικασία ένταξή τη. Προ την ένταξη έστω. Είναι σημαντικό να κινηθεί λοιπόν σε αυτό το δρόμο για την αξιοπιστία μας στην ευρύτερη περιοχή ω κάποιο που προσωπικώ αναμίχθηκε στα πολιτικά πράγματα τη χώρα και ασχολήθηκα με τα πολιτικά πράγματα τη χώρα επί χρόνια, να επιβεβαιώσω ότι το κλίμα στα πολιτικά, ε, στις πολιτικές υποθέσεις της Αλβανίας έχει ε, προχωρήσει. Βεβαίω, η πόλωση είναι ακόμα έντονη, όμως η ατμόσφαιρα έχει βελτιωθεί. Πολλά πολιτικά ζητήματα έχουν επιστρέψει και συζητώνται στην ε, ε, Βουλή της χώρας και οι πολίτες ανταποκρίνονται στο δημοκρατικό διάλογο υψηλών προτύπων, ακόμη και η μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου. Είναι μια βαθιά και ε, εντατική μεταρρύθμιση που χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει από το μια στιγμή στην άλλη. Η υλοποίηση μια τέτοια μεταρρύθμιση χρειάζεται χρόνο. Και εδώ θα ήθελα να αφήσω κατά μέρο την ιδιότητά μου ω ε, ε, Ευρωβουλευτή, αλλά να πω ότι η ΕΕΔ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσαν μεγάλη συνδρομή και βοήθεια στην μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου στην Αλβανία και μπράβο τους. Εδώ να ε, ευχαριστήσω τον εισηγητή που σωστά ε, υποδεικνύει σε ποιου τομεί πρέπει να γίνει πρόοδο. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, δεν έχω κάτι να προσθέσω και για την πολιτική διεύρυνση και την διαδικασία ένταξη βάση ερεσιμότητα. Αυτό ο δρόμο έχει δύο κατευθύνσει. Δεν μπορούμε να γίνουμε όμοιροι πολιτικών χειρισμών. Εάν οι προϋποθέσεις τηρούνται, πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Ιδάλω, παίζουμε με την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ισχύει και για την Αλβανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Έντουαρτ Κούκαν. Ο κύριο Σόλτε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση σε έξι σελίδες. Υποστηρίζουμε σχεδόν όλα τα σημεία στα οποία στέκεται ε, και αναφέρεται, αλλά σε αυτή τη φάση ένα μόνο σχόλιο για την παράγραφο 28. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι σε προστατευόμενη περιοχή υπάρχει οικοδόμηση υδροελεκτρικού εργοστασίου, εργοστασίου παραγωγής υδροελεκτρικής ενέργειας, και αυτό είναι κάτι που καταδικάζουμε, αλλά ε, Βεβαίω είναι απαράδεκτο από τη μια να υπάρχουν έργα σε προστατευόμενε περιοχέ και πρέπει να επαναλάβουμε την έκκλησή μα για προστασία τη βιοπικιλότητα και των εθνικών πάρκων και δρυμών γύρω από γύρω από τον ποταμό αυτό και τις ε, κοιλάδες από που περνάει με τους παραποτάμους του. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα αξίας χιλιάδων ευρώ που για πολιτικούς λόγους σίγουρα αποτελούν ελκυστικές επενδύσεις, ιδίως για δημόσιες ε, ε τράπεζες, όπως η Τράπεζα της Αλβανίας ε, και η Τράπεζα Επενδύσεων. Όμως δεν υπάρχει λόγος να γίνονται επενδύσεις σε χώρους όπου δεν προβλέπεται κοινωνική και οικονομική ωφέλεια, ιδίως σε προστατευόμενες. Ευχαριστούμε ο κύριος Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε προσωπικά και τον κύριο Φλαγκενστάι για τη δουλειά που κάνει. Εγώ ως σκιώδης εισηγητής θεωρώ ότι με μια καλή συνεργασία μπορούμε να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα που να ωφελεί την Αλβανία, η οποία έχει κάνει βήματα, ωστόσο χρειάζεται ακόμη να γίνουν πολλά για να επιταχυνθεί η ενταξιακή διαδικασία. Πρώτα απ' όλα στο σεβασμό και η τήρηση των κριτηρίων της Κοπενχάγης που αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για κάθε κράτος που επιθυμεί να ενταχθεί. Ο πολιτικός διάλογος και μια υγιής δημοκρατία που θα σέβεται την αντίθετη άποψη αλλά και ταυτόχρονα τους νόμους και τις διαδικασίες. Είναι που αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεγονότα όμως όπως αυτά του περασμένου Δεκεμβρίου στο Κοινοβούλιο της χώρας δεν τιμούν κανένα και σίγουρα δεν συνάδουν με κράτος που θέλει να ενταχθεί. Επίσης, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι άλλο μεγάλο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει την Αλβανία. Το οργανωμένο έγκλημα, η σωματεμπορία, η διακίνηση ναρκωτικών είναι τομεί που η Αλβανία χρειάζεται άμεσα να λάβει μέτρα. Επίση, η ελευθερία τη έκφραση, η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωση και των δημοσιογράφων. Η Αλβανία χρειάζεται ακόμα να κάνει βήματα στον τομέα του σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διακρίσει και ο κοινωνικό αποκλεισμό. Η προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των μειονοτήτων Θέλουμε μια Αλβανία η οποία να συνεργάζεται με τους γείτονές της σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Μια Αλβανία η οποία θα τηρεί τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της. Σε αυτό το κλίμα θα πρέπει να επιδιωχθεί η επίλυση προβλημάτων και εδαφικών διεκδικήσεων με τα γειτονικά κράτη, όπως προέτρεψε και ο πρόεδρος Γιούγκερ στην επίσκεψή του τον Φεβρουάριο. Κλείνω λέγοντας ότι μέσα από τις τροπολογίες ελπίζομαι ότι θα κυλήσουν τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η απόφαση του Συμβουλίου για να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της ε, Αλβανίας θα πρέπει να λάβει υπόψη Ορισμένε παραμέτρους που αναφέρονται και στην έκθεση, ανέφεραν και οι προλαλήσαντε συνάδελφοι. Εγώ θα επικεντρώσω το ενδιαφέρον σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι εσωτερικά η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίω τη ελληνική μειονότητα, η οποία είναι η πολυπληθέστερη μειονότητα τη Αλβανία, Έχουν αναφερθεί εδώ πολλά, πολλές παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων και όσον αφορά την καταπάτηση ιδιοκτησιακού καθεστώς, την προσπάθεια μειώσεως ε, του μεγέθους της μειώνοντας με διάφορες μεθόδους νομικιστικές, ε, γκρέμισμα εκκλησιών, ε, καταπάτηση περιουσιών κυρίως σε περιοχές παραθαλάσσιες και πώληση αυτών των διοκτησιών είτε σε οργανωμένο έγκλημα είτε σε ξένες εταιρείε. Και το δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να επισημαθεί είναι η τάση που έχει η Αλβανία να έχει επεκτατικές βλέπεις στα γειτονικά κράτη. Εάν επιληθούν αυτά τα προβλήματα, όλα τα υπόλοιπα σε κάποια στιγμή θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και η Αλβανία να γίνει ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Επιτίδιο. Κύριος Μποστινάρο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, να θυμόμαστε ποιο είναι το σημείο εκκίνησης το 2014 κάθε φορά που συζητάμε για την Αλβανία και πόσο επίμαχες ήταν οι συζητήσεις που γινόντουσαν για την Αλβανία και πόσο σκληρός ήταν ο αγώνας μεταξύ δύο ομάδων συνήθω σοσιαλιστών από τη μια και έλκα από την άλλη. Τώρα, χάρη στον Κνούτ, φαίνεται ότι καταλήγουμε σε μια μάλλον συνενετική έκθεση. Κάτι το οποίο είναι αξιόπαινο και δείχνει και τι πρόοδο έχει πετύχει η Αλβανία οι Αλβανοί θα πρέπει να είναι περήφανοι για την πρόοδο αυτή που πέτυχαν. Εξού και στηρίζω απόλυτα την έκκληση προς το Συμβούλιο να προσφέρει την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Αλβανία. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την ευθυγράμμιση της Αλβανίας με την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εντυπωσιακό και αποτελεί και παράδειγμα για άλλους να κάνουν το ίδιο. Συγχρόνως πρέπει να σημειώσω τον μεγάλο θετικό ρόλο που έχει παίξει η Αλβανία. Το έχουν πει και τα μέσα ενημέρωση που δεν είναι πάντα φιλικά. Τι καλό ρόλο έχει παίξει ο Πρωθυπουργό δηλαδή στην περιοχή. Τέλος, Πρόεδρε, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταφέραμε να πετύχουμε πρόοδο στην Αλβανία χάρη στην σοφή συνεργασία μεταξύ των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την πολύ σοφή απόφαση να σταματήσουμε να τα βάζουμε ένας με τον άλλον είτε πρόκειται για την Αλβανία, είτε για τη Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, διορθώνει ο μιλητής. Για άλλη μια φορά λοιπόν, Πρόεδρε, θέλω να κάνω έκκληση στους συναδέρφους να συνεχίσουμε στην ίδια γραμμή. Γιατί να έχουμε άλλη μια περίπτωση τώρα όπου πρέπει να πούμε στους εταίρους μας, στα κόμματά μας, στην περιοχή, τα αδερφά, τι έχουμε πετύχει. Τέλος, Βόρεια Μακεδονία. Πρέπει να πούμε στους συναδέρφους και τους φίλους από τα αντίστοιχα κόμματα ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να ξεπεραστούν ποτέ και αν ξεπεραστούν τότε θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από τις δικές μας πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρο. Η κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φραγκεστάιν, θεωρώ ότι έχετε παρουσιάσει μια ισορροπημένη έκθεση όσον αφορά το θέμα της ε, Αλβανίας. Ωστόσο, μια και μιλάμε για προαπαιτούμενα, θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε ένα από αυτά που αφορά στην έκθεση και αφορά στον πλήρη σεβασμό των μειονοτήτων, όπω αναφέρθηκε προηγουμένω και από συναδέλφου. Όπω πολύ σωστά αναφέρεται και στην έκθεση, η Αλβανία θα πρέπει να εργαστεί όπω οφείλει για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωση, τη εκπαίδευση, τη αύξηση του αριθμού και των ποσοστών τη απασχόληση των μειονοτήτων ε, στη χώρα, Όμω, ενώ αναφέρεστε σε άλλε μειονότητε, παραδείγματο χάρη των Ρωμάτων, των Αιγυπτίων κλπ., δεν αναφέρεστε καθόλου στη μεγαλύτερη μειονότητα που είναι και η ελληνική. Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζω ότι η Αλβανία ψήφισε πέρυσι νόμο ε, πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όμω αντί να διασφαλίζει αυτό ο νόμο τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη χώρα βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων, διονύζει τι αυθαιρεσίε του προηγούμενου καθεστώτο Χότζα. Είναι ένα βήμα μπροστά για τι υπαρκτέ και τι ανύπαρκτε και κάνει ένα βήμα πίσω για την ελληνική μειονότητα, για την οποία παραμένουν τα εμπόδια στο δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού και ταυτοποίηση των μελών τη, στη δυνατότητα χρήση ελληνική γλώσσα στη δημόσια ζωή, στη δυνατότητα εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, ενώ επίση αφήνεται άλυτο το περιουσιακό. Συνεχίζουν να μην αναγνωρίζονται ω μειωτικέ περιοχέ με πολυπληθέ ελληνικέ κοινότητε, όπω είναι η Χιμάρα, τα ελληνικά χωριά στον Αυλώνα κλπ. Και τα επισημαίνω αυτά γιατί είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε ασφαλώ τα περιστατικά που τα ανέφερε πάλι συνάδελφο προηγουμένω που είχαν προηγηθεί την προηγούμενη χρονιά κατά των ιδιοκτησιών μελών των, ε, τη ελληνική κοινότητα, παραβιάζοντα τα διεθνώ αναγνωρισμένα δικαιώματα των ε, μειονοτήτων και πρέπει να επισημάνω επίση ότι η αλβανική κυβέρνηση πρόθεσε μέτρα καταστροφή των περιουσιών των μελών τη ελληνική εθνική μειονότητα στο πλαίσιο πολιτική ξεριζωμού που εφαρμόζει τη ιστορική παρουσία του ελληνισμού στην περιοχή τη Χιμάρα και παρά τι αρνητικέ συστάσει που έχουν γίνει από, την, από τον συνήγορο του πολίτη τη Αλβανία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κανένας άλλο το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Ρουίθ Καλαβέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να σας πω όσον αφορά τον περιορισμό των σελίδων που λέτε ότι δεν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα έχετε όριο. Ε, έχουμε με τις εσωτερικές μας υπηρεσίες, σε πάση περιπτώσει. Όντω είναι εκτενή η εκθεσή μα, αλλά δεν έχει σημασία ο αριθμό των σελίδων. Αλλά να υπάρχει ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τα μηνύματά μας προς τις χώρες αυτές. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και τον κύριο Φλάγκενστέιν για το σχέδιο εκθεσή του. Εκτιμώ όλος ιδιαίτερω την σαφή του στήριξη και του Ευρωπαϊκού Γενοβουλίου γενικώ που είναι θετικό ε, και είναι υπέρ ε, του βήματο αυτού της Ευρωπαϊκή Επιτροπής να προτείνει το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων με την Αλβανία. Θα ήθελα πάντω να επαναλάβω ότι το καθεστώ υποψήφιας ε, χώρας δόθηκε στην Αλβανία από το 2014 και έκτοτε έχει κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις η χώρα με σταθερή πρόοδο σε διαφορούς τομεί που έχουν να κάνουν με τι πέντε προτεραιότητέ μα. Και γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η σύσταση αυτή είναι βάσιμη και τη στηρίζουμε βέβαια. Επίσης θέλω να πω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η πρόοδος πρέπει να προχωρήσει, να παγιωθεί και γι' αυτό και εκτιμούμε ιδιαίτερος ότι το σχέδιο κειμένου αναφέρει πολλές συστάσεις που πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμες και θα έχουν επιπτώσεις στην εσωτερική συζήτηση στην Αλβανία. Θέλω να αναφέρω τώρα κάποιου ε, τομεί που εκτιμούμε ιδιαίτερω. Για παράδειγμα, δικαιοσύνη, αξιολόγηση. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημαντικό ρόλο διότι έχουμε το καθεστώς του παρατηρητή. Λέτε επίσης να συνεχιστεί ο πολιτικός διάλογος μεταξύ όλων των ε, πλευρών για την μεταρρύθμιση. Ε, πρόοδο στο κράτος δικαίου και την δικαιοσύνη, κυρίως την αντιμετώπιση της διαφοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Μιλάτε επίσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα και μειονοτήτων, αλλά και να διασφαλίσουμε και την εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία της ιδιοκτησίας. Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο όσον αφορά επίσης την νεολαία. και έτσι να γίνουν οι αλλαγέ που χρειάζονται υπέρ της συμφιλίωσης. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φλάκενστάιν και βέβαια και όλα τα μέλη της Επιτροπής σας και όλους τους ευρωβουλευτές που βοήθησαν για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Κνούτ Φλάκενστάιν. Βεβαίως, βεβαίως, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Νομίζω ότι υπόθηκαν όλα. Σύντομα θα καταλήξουμε πιστεύω σε ένα κοινά αποδεκτό κείμενο και ελπίζω το Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα να είναι εξίσου ομόφωνο και σαφές. Ευχαριστώ Κνούτ για τη συντομία της παρουσίασης. Τώρα, χρονοδιάγραμμα. Όπως και για τη Σερβία και το Κοσφοπέδιο. Οπότε, 30 Αυγούστου, 11 ώρα για τροπολογίες. Αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν κλείσουμε για το πρωί, σας πενθυμίζω. και μέτρησα. Από τα πάνω από 70 μέλη της Επιτροπής μας, μόνο 7 είναι παρανόντες. Και οι 7 βεβαίως είναι υπέροχοι γιατί έμειναν μέχρι τέλους. Αλλά παρακαλώ να πείτε στους συναδέλφους σας ότι έχουμε κοινή συνάντηση με τη ΛΥΜΠΕ στο PHS 3 σε 50 στις 2.30 μέχρι τις 3.30 και κατόπιν έχουμε ένα διαβριμένο προεδρείο ε, και κλεισμένων από τις 3.30 μέχρι τις 4.30 ως προετοιμασία για τη συνάντηση με την κυρία Μογκερίνη και μετά από τις 4.30 μέχρι τις 5.30 θα έχουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικό, Εξωτερικών του Ιράν σε αυτή την αίθουσα. 4.30 με 5.30 αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Όλα αυτά έχουν ε, αποσταλεί. Και αύριο θα έχουμε ένα επιπλέον θέμα στη μέση διάταξη, κατάσταση στην Μολδαβία, συγκεκριμένα στο Κισινάου. Καλή όρεξη σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή ζήτηση, για τη Σερβία, το Κοσμοπέδιο και την Αλβανία.